So, I think we Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την απογευματινή συνεδρίαση. Έχουμε μια κοινή συζήτηση για δύο πράξεις κάτω εξουσιοδότηση. Να σας υπενθυμίσω το ιστορικό μετά από την τεχνική συνεδρία των πολιτικών συμβούλων στις 11 Νοεμβρίου. Έχουμε σήμερα την παρουσίαση τον κύριο Ολιβιέ Ονιντή, αναπληρωματικό διευθυντή, γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών. Η μία φορά το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ε, και το άλλο αφορά το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης. Η Κομισιόν παρουσίασε μια πρόταση τον Οκτώβριο και υπάρχει μια προθυμία δύο μηνών για αντιρρήσεις. Οι δύο πράξεις κατά ακολουθούν επειδή το Κοινοβούλιο στην προηγούμενη θητή έχει εκφράσει αντίρρηση σε δύο παρόμοιες πράξεις κατά Στην περίπτωση της πράξης για το Ταμείο Ασφαλείας περιλαμβάνεται μια συγκεκριμένη δράση, συγκεκριμένα οι δράσει ελέγχου των συνόρων, όπως μέτρα ελέγχου και εποπτείας των συνόρων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν υψηλές ή δυσανάλογες μεταναστευτικές πιέσεις, περιοχές hot spot και στήριξη τέτοιων δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες. Όσον αφορά την πράξη κατεξιοδότησης για το Ταμείο Σύλλου μετανάστευση και Ένταξης. Ε, έχουμε μια νέα δραστηριότητα η οποία αφορά τις εγκαταστάσεις υποδοχής και κράτησης για παρατύπω διαμένοντε υπηκόους τριτών χωρών ή αιτούντε άσυλο σε χώρες που αντιμετωπίζουν υψηλή ή δυσανάλογη μεταναστευτική πίεση. Τι έγινε λοιπόν με αυτά. Φαίνεται ότι το Κοινοβούλιο δεν είχε ενημερωθεί για τη σύνταξη των δύο αυτών πράξεων κάτω εξουσιοδότηση. Πολλές πολιτικές ομάδες, σοσιαλδημοκράτε, γκουε, πράσινοι, ρινιού, ζήτησαν από την Επιτροπή μας, ζήτησαν η Επιτροπή μας να ενημερωθεί για το ιστορικό και τα βασικά στοιχεία και την διαδικασία λήψης αποφάσεων η Κομισιόν αναγνώρισε εκ των υστέρων γραπτός πως είχε υπάρξει μια παράληψη ε, ενημέρωση του Κοινοβουλίου και ότι λυπόταν γι' αυτό. Καλωσορίζουμε λοιπόν τη συμμετοχή της Κομισιόν στην ανταλλαγή αυτή απόψεων ε, και το ότι αναγνώρισε το πρόβλημα αυτό. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να τονίσω ότι η έλλειψη των σχετικών ε, πληροφοριών ε, συγκεκριμένα το ότι δεν εστάλει το σχέδιο των πράξεων αυτών αντιβαίνει το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να ενημερώνεται για πράξη κατά εξοδότηση όπως αυτό έχει καταγραφεί στην ε, Διοργανική Συμφωνία περί καλύτερης νομοθεσίας του 2016 σύμφωνα με την οποία Συμβούλιο και Κοινοβούλιο θα λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους ε, εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Επίσης, τίθεται ένα αμφιβόλο το δικαίωμα εξέτασης ε, του Κοινοβουλίου και θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε παράταση των προθεσμιών έτσι ώστε το Κοινοβούλιο ή οι βουλευτές να έχουν δικαίωμα να ασκήσουν το ε, λόγο δικαίωμα. Υπενθυμίζω ότι οι δύο αυτές πράξεις συνδέονται με δύο προηγούμενες ε, κατεξοδότηση πράξεις για τις οποίες είχε γύρει αντίρρηση η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου στην προηγούμενη θητεία γιατί υπήρχε η έννοια των ενεχόμενων κέντρων για τα οποία δεν υπήρχε νομική βάση ή εξήγηση για το τι ακριβώς σημαίνει. Οπότε, αφού υπενθυμίσαμε το ιστορικό της υπόθεσης, θα δώσω τώρα τον λόγο στον διακεκριμένο μιλτή μας, τον κύριο Ολιβιέ ONID από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής. Έχει τον λόγο για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να έρθω εδώ και να σας εξηγήσω το σκεπτικό για τις προτάσεις αυτές. Είχατε κι εσείς ε, μια πολύ έτσι, αναλυτική εισαγωγή. Ε, σημειώνω και εγώ. Έχουμε κάνει λάθη πράγματι και ζητούμε συγγνώμη. Και σίγουρα μας ενδιαφέρει και εμάς να ενημερώνεστε εσείς όσο πιο νωρίς γίνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας. Για να υπάρξει η δική σας εποπτεία σε οποιαδήποτε μελλοντική πράξη. Μας είπατε ότι οι δύο αυτές πράξεις κατατίθεται πολύ αργά διότι δυστυχώς στην προηγούμενη θητεία κατά το τέλος της ε, απορρίψατε δύο πολύ παρόμοιες πράξεις που περιείχαν ακριβώς την ατυχή έκφραση Control Center, ελεγχόμενο κέντρο. Και αυτό σας δημιουργούσε προβλήματα. Μάλλον ήταν καλή τελικά η κίνησή σας, γιατί μας έχουν ξεπεράσει τα γεγονότα και δεν είναι πλέον το βασικό μας μέλημα αυτά τα κέντρα. Και έχουμε πλέον περάσει κάτι διαφορετικό. Είμαστε σε ένα άλλο τρένο τώρα. Λίγη η χρηματοδοτική αυτή περίοδος, έχουμε διαθέσιμα κονδύλια Δυστυχώς όμως υπάρχουν αρκετά κράτη-μέλη που χρήζουν περαιτέρω υποστήριξης. Κυρίως για να βελτιωθούν οι συνθήκες στα κέντρα υποδοχής, αλλά και για να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες πιέσεις σε ορισμένα σύνορα. Με διάφορους τρόπους, κλίονες, του ενός μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτή την χρηματοοικονομική υποστήριξη. Αυτό όμως το οποίο προτείνουμε είναι να προχωρήσουμε με αυτές τις τροποποιημένες κατεξουσιοδότησιν πράξεις. Γιατί από δημοσιονομικής πλευράς αυτό είναι ο πλέον ε, διαφανής, ε, καθαρός, αν μπορώ να το πω έτσι, τρόπος για να προχωρήσουμε. Δύο εναλλακτικέ υπάρχουν ουσιαστικά. Να χρησιμοποιήσουμε τα ταμεκτάκτη της ανάγκης, αλλά τα έχουμε τεντώσει μέχρι εκεί που ετοιμάζεται να σπάσει το σκηνή αυτά τα ταμεία και χρειάζεται πραγματικά μεγάλη πειθαρχία για να περιορίσουμε τη χρήση αυτών των κονδυλίων έκτακτη ανάγκη στα απολύτω αναγκαία. Όταν δηλαδή μιλάμε για πραγματικά κάτι κατεπήγον, λίγος χρόνος μας μένει για να προγραμματίσουμε τη χρηματοδότηση και η άλλη εναλλακτική είναι να αναθεωρήσουμε ε, σε βάθος τις εθνικές ε, κατανομές ε, κονδυλίων, τα εθνικά κονδύλια. Αυτό βέβαια θα ανοίξει την πόρτα ε, σε αξιώσεις ε, και διεκδικήσεις από όλα τα κράτη-μέλη, οπότε δεν θα μπορέσουμε να μείνουμε σε αυτή τη στοχευμένη υποστήριξη που θέλουμε να παρέχουμε, δηλαδή κέντρα υποδοχής αφενός και διαχείριση πιέσεων σε ορισμένα σύνορα αφετέρου. Αυτές είναι οι δύο προτεραιότητες, οι δύο τομείς στο οποίες στοχεύουμε. Ακούσαμε τη θέση και τη σημειώνουμε, τη θέση του Κοινοβουλίου ε, στην προηγούμενη μας προσπάθεια. Δηλαδή, άρα τα ελεγχόμενα αυτά κέντρα δεν περιλαμβάνονται πια στο κείμενο. Και έτσι περιοριζόμαστε στο πεδίο παρέμβασης ε, για τα κέντρα υποδοχής, όπως σας είπα, και τη διαχείριση των συνόρων. Ευχαριστώ. Thank σας ευχαριστώ πολύ κύριο Ονιντή. Κανονικά σε αυτό το σημείο θα έπρεπε να έχουμε ένα γύρο από τους συντονιστές και εν συνεχεία θα έπαιρναν το λόγο οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Όμως δεν βλέπω κάποιον ασυντονιστή από το ΕΛΚΑ, άρα ε, επόμενος θα ήταν ο συντονιστής από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, η δηλαδή, Μπίρκη Τσίπελ. Πριν όμως πάρω εγώ το λόγο, ίσως καλύτερα θα ήταν να τον δώσω σε έναν άλλο συντονιστή που είναι παρόν και συγκεκριμένα η συνάδελφος ε, την Καστρίκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Κομισιόν που μας ε, κατέθεσε αυτές τις προτάσεις. Πράγματι, είχαμε ανησυχίες για αυτή την έννοια του κέντρου ελέγχου ή ελεγχόμενου κέντρου και τώρα μιλάμε για στήριξη για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Κροατίας, αν κατάλαβα καλά, για το Ταμείο Ιστορικής Ασφάλειας ε, και για τη Βουλγαρία και μιλάμε επίσης για στήριξη στο σύστημα ΆΜΙΦ, δηλαδή για το άσυλο μετανάστευση για Ελλάδα ε, σε ό,τι αφορά τις δομές υποδοχής, έτσι. Λοιπόν, έχουμε κάποιες ερωτήσεις και για τις δύο προτάσεις. Όπως γνωρίζετε, ήδη έχουμε και τις ανησυχίες μας για τις πρακτικές στα σύνορα Κροατίας-Βοσνίας. Ε, γίνεται πολλής λόγος και υπάρχουν πολλέ καταγγελίες για αποθήσεις σε αυτή τη μεθόριο. Και αυτό που βλέπουμε επιτόπου είναι ότι οι πρακτικές γίνονται ακόμη πιο ανησυχητικές. Άρα, αντί να διασκεδάζονται ανησυχίε, ε, φαίνεται τα πράγματα να επιδεινώνονται και οι φήμες για το μηχανισμό ε, διέλευσης, ε, το transit mechanism, δεν έχουμε ακόμη κάτι συγκεκριμένο και δεν ξέρω κατά πόσον αυτό συνάδει με την υποχρέωση για διαφάνεια. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε λίγο περισσότερα πράγματα για τα κριτήρια ε, Φερρυπίν που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να χορηγήσει έξτρα για τη διαχείριση συνόρων τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαίωμα στην πρόσβαση λαμβάνονται υπόψη και σε ποιο βαθμό. Το ίδιο ισχύει για το ΆΜΙΦ, για την Ελλάδα. Πρόσφατα, χθε, ακούσαμε ε, ποια είναι τα νέα σχέδια της Ελλάδας να μεταφέρει ε, στην ε, υπηρετική χώρα πολύ κόσμο και να δημιουργήσει κλειστά κέντρα που ουσιαστικά είναι φημισμός γιατί κανονικά θα πρέπει να μιλάμε για κέντρα κράτησης. Όλα αυτά πραγματικά μας ε, ανησυχούν ε, και τι σχέση έχουν όλα αυτά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και το δικαίωμα ασύλου. Άρα το ερώτημά είναι σε ποιο βαθμό Ε, θα ελέγχουμε ε, το πώς δαπανούνται αυτά τα επιπλέον κονδύλια. Πριν από δύο εβδομάδες ε, είχαμε συζητήσει για αυτό το σχέδιο νόμου, το νομοσχέδιο της Ελλάδας και η Κομισιόν είπε ότι θα μελετούσε το κατά πόσον συνάδουν μετά όσον για την, τα περί και θα ήθελα να ακούσω αν εσείς έχετε πλέον κάποια συγκεκριμένα πράγματα να μας πείτε και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτών των κατεξουσιοδότης κανονισμών θα θέλαμε να μπορούμε να ασκήσουμε το δικαίωμα εξέτασης ε, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά θα θέλαμε μία παράταση. Ευχαριστώ. Είχαμε αρκετέ ε, ερωτήσει και παρατηρήσει, θα επανέλθουμε. Εγώ θα μιλήσω στο τέλος. Οπότε ε, για την ώρα έχετε τον λόγο εσείς κύριε Χουκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, ε, τώρα δεν ξέρω αν τα καλούμε κέντρα υποδοχής ή κάτι διαφορετικό. Αυτά θα τα ε, διαχειρίζονται οι αρχές των κρατών μελών ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν τα λειτουργούν τα κράτη-μέλη, όπως αυτή τη στιγμή θα υπάρχουν κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές ε, που η Κομισιόν ή κάποιος άλλος θα φροντίζει να τίνονται. Παραδείγματο χάρη στη χώρα μου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχαμε κάποιες σκανδαλώδεις ε, συμπεριφορές στο παρελθόν όσον αφορά τα παιδιά τα οποία δεν τα φρόντιζαν σωστά. Και φαντάζομαι και στα άλλα κράτη-μέλη θα υπήρχαν άλλα. Οπότε φαντάζομαι καλό είναι να υπάρχουν κάποια ε, βασικά πράγματα, π.χ. πρόσβαση στα σχολεία. Ε, νομίζω όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση σύμφωνα και με τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και όπου δυνατόν μαζί με τα, παιδιά, τα ντόπια εκεί πέρα να μαθαίνουν την γλώσσα. και επίση θα φροντίζουμε να μην είναι άστεγοι γιατί το καλοκαίρι εγώ πήγα στην περιοχή κοντά στο Καλαίο που χίλιοι πρόσφυγες τώρα δεν υπάρχουν εκεί πέρα οργανωμένες εγκαταστάσεις, κοιμούνται στο δάσος κοντά σε χωματερές. Ε, δεν ξέρω αν ε, υπάρχουν κάποιες σχετικές προδιαγραφές. Επίσης, αν θα πρέπει οι πρόσφυγες να εργάζονται στη χώρα μου, δεν επιτρέπεται, τους απαγορεύεται, κατόπιν είναι βλακώδες. Γιατί συχνά είναι άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν Υπάρχει ένα στο καλέ ο οποίος ε, είναι δάσκαλο μιλάει πέντε γλώσσες. Δεν μπορεί να δουλέψει σε ένα σχολείο. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν έχει κάτι σχετικά. Και τέλος, θετικό αυτό το οποίο είπε η Κομισιόν ότι θέλει ένα νέο σύμφωνο ε, σε 100 μέρες. Είναι κάτι το εντελώς ε, καινούργιο θα βασίζεται στους υφιστάμενου κανονισμού. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επεκτείνουμε λίγο το τεχνικό θέμα της συζήτησής μας και μια που εγώ έχω λίγο πολύ τεχνικές παρατηρήσεις ε, νομίζω καλό είναι να απαντηθούν πρώτα οι ερωτήσεις που έγιναν. Έχετε τον λόγο. Α, συγγνώμη. Δεν σας είδα ε, που σηκώσατε το Νόμιζα ότι είχατε σημειώσει το όνομα, είμαστε εδώ σε αυτή τη γωνία δυστυχώς. Χαίρομαι που συμμετέχω, αλλά λυπούμε κιόλα γιατί είναι πολύ σοβαρή αυτή η συζήτηση και όπως είπατε κυρία Πρόεδρε, η αναθεώρηση αυτών των δύο πράξεων έχει ήδη απορριφθεί από το Κοινοβούλιο και βεβαίω το ότι έχουν φύγει τώρα τα κέντρα ελέγχου και δεν πρέπει να ανησυχούμε δεν ξέρω, εγώ το βρίσκω εκπληκτικό γιατί ανησυχώ ακόμη περισσότερο τώρα, ειδικά δεδομένων των εξελίξεων ε, χτες ε, στην Ελλάδα, γιατί ουσιαστικά αυτό το οποίο λέμε σε σχέση με την πράξη για το Ταμείο Σύλλου και Μετανάστευσης, ε, που μιλάμε για 200 εκατομμύρια ευρώ, στο πλαίσιο του ε, η Κομισιόν αφήνει ανοιχτό το θέμα κέντρων κράτησης είναι πάρα πολύ προβληματικό γιατί ξέρουμε που θα πάνε τα λεφτά αν δούμε τι ανακοίνωσε χτες η Ελλάδα και αν συμφωνήσουμε επιτρέπουμε τα λεφτά του Ευρωπαίου φορολογούμενου να χρηματοδοτήσουν κέντρα κράτησης. Ε, η ελληνική κυβέρνηση το είπε ανοιχτά. Μίλησε για 5 έως 10.000 άτομα που θα μετακινηθούν. Κάποιοι από αυτούς ε, δε σε ακατοίκητα νησιά ε, θα είναι το Γουαντανάμο της Ευρώπης. Ε, δηλαδή ότι το σκέφτονται είναι αδιανόητο και νομίζω ότι ε, είναι αντίθετο με την οδηγία περί επιστροφών που λέει ότι η κράτηση πρέπει να είναι η τελευταία λύση. Λοιπόν, έχω κάποιες ερωτήσεις και κάποιες προτάσεις. Πρώτα απ' όλα πρόθεσή μας είναι να καταθέσουμε μια ένσταση η οποία θα συζητηθεί στην συνεδρίαση των ε, συντονιστών. Σκοπεύουμε δε να ζητήσουμε από την Κομισιόν να μην υπάρχει δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν κέντρα κράτησης και θα ήθελα να σας ζητήσω κυρία Πρόεδρε να ενημερώσετε την Κομισιόν ότι θα ζητήσουμε παράταση της προθεσμίας έτσι ώστε και το Κοινοβούλιο να μπορέσει να εξετάσει Επίσης ε, ζητάμε να υπάρξει μια γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας για την συμβατότητα της πράξης αυτής με τον υφιστάμενο κανονισμό ασύλου και μετανάστευση, ειδικά το εκτιμώντας 38, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, ε, δεν θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή τηρείται. Ε, αυτή είναι λοιπόν η πρότασή μας. τώρα για το άλλο το οποίο αφορά το Ταμείο εσωτερική Ασφαλείας θα είναι τα 63 εκατομμύρια και λένε ότι στο τεχνικό επίπεδο θα πάνε αυτά τα λεφτά σε Κροατία και Βουλγαρία για επιτήρηση των συνόρων. Όχι για επιτήρηση δηλαδή παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά για επιτήρηση και διαχείριση των συνόρων. Ε, και πάλι αυτό είναι συγκλονιστικό δεδομένου του ότι είναι αναφυσβήτητο ότι έχουν λάβει χώρα παραβιάσεις, ειδικά στα κροατικά σύνορα. Αν δείτε το παράδειγμα του περιστατικού της προηγούμενης εβδομάδας, όπου είχαμε βίαιες αποθήσεις και πυροβολισμούς ε, κατά μεταναστών από μία περίπολο στα σύνορα. Ε, διότι ότι αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα για χρηματοδότηση είναι ε, πολύ προβληματικό. Λοιπόν θα πρότεινα να στείλουμε μία επιστολή στην Κομισιόν και να περιλάβει στα κριτήρια επιλεξιμότητας οι χώρες να συμμορφώνονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα στις δραστηριότητες ελέγχου των συνόρων και να ενημερωθούμε αν αυτό περιλαμβάνεται. Και νομίζω ένα αίτημα επίσης ε, προς την Πρόεδρο δεδομένη της ε, συζήτηση ε, των συντονιστών την επόμενη εβδομάδα για να ζητηθεί μια παράταση της προθεσμίας για να μπορέσουμε να ασκήσουμε και εμείς ε, τα ελεκτικά μας καθήκοντα. Σας ευχαριστώ. Όπως είπα, επεκτείνουμε λίγο το τεχνικό πεδίο. Πριν δώσω όμως τον λόγο στον κύριο Ονίδη, να σιγουρευτώ ότι δεν ξέχασα κανέναν. Ωραία. Κύριε Ονίδη, έχετε τον λόγο. Εγώ θα κάνω μια πιο τεχνική παρατήρηση στο τέλος. Ευχαριστώ, αγαπητή Πρόεδρε, κυρία Ζίπελ. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον για τα ευρύτερα ζητήματα και ελπίζω να αναλάβει σύντομα καθήκοντα η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί έτσι θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε και ε, μια πολιτική συζήτηση με τους ε, αρμόδιους επιτρόπους και αντιπροέδρους για το τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να πλαισιωθεί αυτό το νέο ε, σύμφωνο για τη μετανάστευση. Σας κατανοώ και νομίζω ότι όλοι στην ίδια θέση βρισκόμαστε, όλοι περιμένουμε να ξεκινήσουν πραγματικά οι συζητήσεις. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα για όσα σχόλια έγιναν. Καταρχάς, ό,τι αφορά τον κατάλογο των κρατών μελών που δυνητικά θα μπορούσαν να αποφεληθούν οικονομικά από αυτούς τους δύο κατεξιότητες κανονισμούς. Σε ό,τι αφορά το ΆΜΙΦ, έχουμε την Ελλάδα φυσικά, λόγω της κατάστασης πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη χώρα αυτή που υποδέχεται ένα τεράστιο μερίδα μεταναστών στην Ευρώπη. Έχουμε και την Κύπρο που και αυτή δέχεται πιέσεις, τη Βουλγαρία, τη Μάλτα, την Ισπανία, ακόμη και τη Γαλλία. Για το Ταμείο Στήρικης Ασφάλειας και εδώ δεν είναι μόνο η Κροατία, αλλά και η Βουλγαρία, η Ισπανία και η Ελλάδα. Είναι υποψήφιες χώρες για τα επιπλέον αυτά κονδυλάρια. Είναι ευρύτερη λίστα. Τώρα, για το ευρύτερο ζήτημα το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια αυτά, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση, νομίζω πρώτα και πάνω απ' όλα, αν διατεθεί χρηματοδότηση προς τα κράτη-μέλη, αυτό γίνεται ακριβώς για να βελτιωθούν οι συνθήκες. Και πάντοτε βέβαια σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η νομοθεσία και το συνολικό νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αυτά τα κονδύλια δεν πρόκειται να ε, δαπανηθούν ουσιαστικά για να διονυστούν καταστάσεις που θα ήταν παράνομες και δεν θα ευθυγραμμίζονταν με την αξιοπρέπεια, την ατομική αξιοπρέπεια Ακριβώς για το αντίθετο πρόκειται. Ακριβώς επειδή δυστυχώς υπάρχουν κάποιες καταστάσεις ε, που πόρο απέχουν ε, του να είναι βέλτιστες, πρέπει, έχουμε καθήκον και χρέο να στηρίξουμε αυτά τα κράτη-μέλη και οικονομικά μεταξύ άλλων. Έχουμε ένα συνολικό νομοθετικό πλαίσιο όπως γνωρίζετε. Υπάρχει μάλιστα και μια επικαιροποιημένη σύγχρονη πρόταση επιτάπητος ε, για την πτυχή, το σκέλος της υποδοχής. Δυστυχώς στην προηγούμενη νομοθετία δεν καταφέραμε να το εγκρίνουμε, αλλά ελπίζω να τα πάμε ακόμη καλύτερα μέσω του Συμφώνου μετανάστευση. Ό,τι χρηματοδοτείται με ευρωπαϊκά κονδύλια γραμμίζεται απόλυτα και αυτό το ελέγχουμε, το επαληθεύουμε στη φάση της εξέτασης ε, των προτάσεων των κρατών μελών, αλλά και στη διάρκεια ζωής των προγραμμάτων. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο μας δίνει τη δυνατότητα, το κίνητρο, ε, είναι ένας μοχλός ε, ακόμη για να αντιμετωπίσουμε κάποια από τα ζητήματα. Αν θεωρήσουμε και αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν πρακτικές σε ορισμένα κρατημέλη στους τομείς αυτούς, διαχείριση συνόρων, υποδοχή, που δεν εφηγραμμίζονται με τα δέοντα ε, και για τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι αφορά τι αποθήσει. σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση που γίνεται με βάση τις έρευνες. Σίγουρα δεν είναι διαφανής και συμφωνώ μαζί σας και ελπίζω πολύ σύντομα να μπορέσουμε να σας δώσουμε πρόσθετες πληροφορίες. Είμαι και διατεθμένος να ξανάρθω στην Επιτροπή σας ε, και να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες ε, για τα πορίσματα αυτών των ε, ερευνών. συνεργαζόμαστε με ανεξάρτητες οργανώσεις ε, ή πατή αρμοστή για τους πρόσφυγες, το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό, βοηθάει σε αυτές τις έρευνες και θα παρασχεθεί ε, αυτή η δυνητική βοήθεια που θα αποτελέσει και αυτή έναν ακόμη μοχλό για να ασκήσουμε πίεση και να ζητήσουμε ε, να γίνονται ε, τα πράγματα όπως πρέπει και να μην υπάρχει αυτού του κακοδιαχείριση που βλέπουμε στην βοσνοκρατική μεθόριο. Άρα θα υπάρχουν ευθύνες για τα κράτη που δεν ε, τηρούν τους κανόνες. Αυτά που είπατε για τα πρότυπα ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι, πράγματι, κάποια πρότυπα, κάποιοι κανόνες είναι ενσωματωμένοι στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε ό,τι αφορά ε, τώρα το χρηματοοικονομικό επίπεδο υπάρχουν ε, και εκεί πράγματα πρέπει να λάβουν υπόψη. Υπάρχουν ε, τα ελάχιστα πρότυπα. δεν μπορώ εγώ να επηρεάσω τα, τις προδιαγραφές των κέντρων υποδοχής, για παράδειγμα, αλλά μπορώ σίγουρα να ασκήσω πίεση περισσότερη σε ό,τι αφορά τον έλεγχο δηλαδή, να εντείνουμε τους ελέγχους. Μόνο που δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτά τα εργαλεία για αυτό το σκόπο. Μπορώ, επαναλαμβάνω, να ασκήσω περισσότερο έλεγχο. Για το νέο αυτό ελληνικό νομοσχέδιο και νόμο η αξιολόγηση μας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη για τον πολύ απλό λόγο πως έχουμε μια διαδραστική συζήτηση με την ελληνική κυβέρνηση, με τις ελληνικές αρχές ώστε ήδη από τώρα να επιτευχθούν κάποιες βελτιώσεις. Πάντως, ακόμη περιδές πρόκειται. Δεν είναι μια πρόταση που έχει κατατεθεί επίση με δημιουργία κλειστών κέντρων θα την αναλύσουμε, δεν είχαμε γνώση, θα αναλύσουμε την ιδέα προς το παρόν αυτή με τη δέωσα σοβαρότητα ε, και ενδελεχώς και βεβαίως και θα επανέλθουμε, είμαστε τεθειμένοι πολύ γρήγορα να επανέλθουμε και να σας δώσουμε ε, τις τελευταίες μας πληροφορίες και την ανάλυση μας ε, για τους δύο μήνες. Δικό σας δικαίωμα είναι και αν θέλετε αυτή την παράταση μπορείτε να μας ενημερώσετε, αλλά καλό θα ήταν να μην καθυστερήσει πολύ να δοθεί αυτή η χρηματοδότηση. Πρέπει να δοθούν τα κονδύλια για του χρόνου, αλλιώς θα χαθούν, πολύ απλά. Και σας παρακαλώ να μην θεωρήσετε ότι είναι ανταμοιβή αυτά τα κονδύλια, ε, εντό αγωγικών ανταμοιβή, προ κράτη-μέλη που δεν τα κάνουν τα πράγματα όπως πρέπει, δείτε το ω κίνητρο. Ω κίνητρο για τη βελτίωση των συνθήκων υποδοχή και διαχείριση των συνόρων. για αυτό το πολύ σοβαρό δυστυχώ, ακόμη φαινόμενο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Thank Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στον συντονιστή των σοσιαλιστών διότι ήθελα να κάνει κάποιες ε, γενικότερες και πιο τεχνικές ε, παρατηρήσεις. Όμως παρατήρησα ότι και ο συνάδελφος Αβραμίδη πρέπει, θέλει να, Αρβανίτης με συγχωρείτε, θέλει κάτι να προσθέσει στη συζήτηση. Ε, εκτιμώ τη συγγνώμη, αλλά ξανά και ξανά βλέπουμε διάφορες μορφές μη σεβασμού της, χρήσης, της αγαστής συνεργασίας μεταξύ των θεσμών και ως εισηγήτρια για τις, ε, τα αποδεικτικά στοιχεία να σας πω ότι μόλις αυτές τις μέρες παρατήρησα μια μη διαφανή συμπεριφορά όχι μόνο από πλευρά της DG Home και ίσως αυτό να είναι κάτι που θα πρέπει να το αξιολογήσουμε με την Επιτροπή. Όμως ε, όπως έλεγε σαφώς ο κύριος ε, Νίλη και το τόνισε μάλιστα. Ίσως θα πρέπει το Κοινοβούλιο να συμμετέχει όσο γίνεται πιο γρήγορα και αυτό έτσι ώστε να αποφευθεί ότι τελικά να μπορούμε απλά να δεχτούμε ή να απορρίψουμε μια πρόταση ανάλογα, μάλλον σε σχέση με τις ε, ε, κατά εξουσιοδότηση πράξης. Ίσως θα μπορούσατε και να στείλετε σχέδιο αυτής ε, κάθε φορά εγκαίρω, ώστε να προειδοποιηθεί η Κομισιόν και να μπορεί να διορθώσει τα προβλήματα ενδεχόμενα πριν να τα εγκρίνουμε ε, εμείς ατύπως. Αυτό λοιπόν θα μπορούσατε ίσως να το λάβετε υπόψη τώρα αλλά και για τη νέα Επιτροπή. Αυτά λοιπόν για τις ε, διάφορες διαδικασίες, αλλά τώρα και ο κύριος Σερβανίτης θέλει να προσθέσει κάτι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Που μου δίνετε το λόγο, εκτός που ε, δεν είχα το δικαίωμα, δεν μιλάμε για... Please. Συμπληρώνω στις εισηγήσεις των δύο ε, συναδέλφων. Δεν μιλάμε για, πολι... για ανθρώπους που θα πάνε στην ενδοχώρα. Πηγαίνετε στο Google Earth και βρείτε το νησί Λεβίθα. Είναι ξερονήσι. Θα επιτρέψουμε, θα δώσουμε χρήματα για να κάνουμε στην Ευρώπη σε ξερονίστια κέντρα κλειστού ή ανοιχτού, κλειστού λέτε εσείς, τύπου. Γκουαντάναμο στην ε, Ευρώπη. Αυτό το ανακοίνωσε χθε η ελληνική κυβέρνηση. Εμεί βγάλαμε δελτίο τύπου, θα καταθέσουμε σχετική ερώτηση βεβαίω στην Κομισιόν και θα ενημερώσουμε το Σώμα. Ήθελα αυτή τη μικρή, πολύ σημαντική για μένα επισήμανση να το μάθουν οι συναδελφοί μου εδώ στη Λίμπε. Just Σας ευχαριστώ. Ε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να χρησιμοποιηθεί ε, η χρηματοδότηση αυτή, αν το στηρίξετε βεβαίως, ε, πλήρως με το υφιστάμενο ευρωπαϊκό δίκαιο αλλά και με κάποια από τα στοιχεία που είναι αυτή τη στιγμή επιτάπητο στις ε, διάφορες προτάσεις ε, ειδικά αυτή για την υποδοχή. Η δεύτερη πτυχή προς την κυρία Τσίπελ δεν υπήρχε κάποια πρόθεση να παρακάμψουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ειδικά αφού την προηγούμενη φορά αντιμετωπίσαμε άρνηση, γιατί δεν σας είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως. Οπότε δεν ε, είναι η δική μου η θέση των πολιτικών προϊσταμένων μου να δεσμευτούμε επισήμως. Αυτό το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω εγώ στο επίπεδό μου ε, είναι για αυτό εδώ, είναι ότι τακτικά θα ενημερώνουμε για τη χρήση αυτών των κονδυλίων αλλά και για μελλοντικές πράξεις κατεξιοδότηση θα κάνουμε τα απαραίτητα βήματα για να ενημερώνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συγκεκριμένα την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ εγκαίρως. Ε, είστε σύμμαχός μας, ε, ξέρετε αυτά, σε αυτά τα θέματα είστε σύμμαχός μας. Okay, at least I think that's... Ε, μάλιστα, νομίζω ότι τουλάχιστον αυτή η δήλωση για το μέλλον, για τα ζητήματα τα οποία είναι πιο ουσίας, αφορά και την ε, συζήτηση για τη νέα Κομισιόν για το νέο μεταναστευτικό σύμφωνο όπως ε, λένε και είναι Κομισιόν. Ελπίζω να ακολουθήσει αυτό το οποία λέει το Κοινοβούλιο και όχι απλά να ε, πάει στα κράτη-μέλη. Ελπίζω λοιπόν να γίνει μια νέα αρχή. Κάποιες προτάσεις έχουν γίνει στην διαδικασία αυτή και βεβαίως όπως ε, επισημάναμε αυτό θα πάει στην συνεδρίαση των συντονιστών αρχές Δεκεμβρίου. Και ειδικά το θέμα αυτό της παράτασης ε, ή όχι. Ε, λοιπόν, έχει παραταθεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, οπότε θα συνεδριάσουν οι συντονιστέ πολύ πιο πριν και μπορούμε να λάβουμε μια σωστή απόφαση για τα αιτήματα αυτά τα σημερινά. Τούτου λεχθέντος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους, να ευχαριστήσω και τον κύριο Ονιντή που ήρθε εδώ και ήταν στη διάθεσή μας αμέσω να απαντήσει στις ερωτήσεις και να εξηγήσει τι υπάρχει πίσω από αυτή την πρόταση. Οπότε συνάδελφοι, Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Λοιπόν, ξεκινάμε τρία λεπτά νωρίτερα, αλλά καλό είναι να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε το επόμενο σημείο στην ημερήσια μας διάταξη, που μιλά για το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μετανάστευσης από τις παγκόσμιες τις τοπικές κυβερνήσεις να καλωσορίσω όσους βρίσκονται εδώ στο Προεδρείο, ορισμένοι παλιότεροι συνάδελφοι θα θυμούνται ίσως ότι έχει γίνει παράδοση να καλούμε τους ε, συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Μετανάστευση για να παρουσιάζουν την έκθεσή τους, εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών καθώς και των ε, κυβερνήσεων ανά το κόσμο και είναι πολύ σημαντικό σημείο αυτό για ε, την ε, αντιμετώπιση του θέματος τώρα. Αυτή τη φορά, αν έχω ενημερωθεί σωστά, ε, η έκθεση, το θέμα, όπως είπα, ήταν από την παγκόσμια συντοπική ε, διακυβέρνηση, ο ρόλος των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών ε, για την εξασφάλιση ασφαλών δρόμων. Είναι σχετικό με διάφορους φακέλους που αφορούν τη μεταρρύθμιση Ε, των ε, νέων ειδών μετανάστευσης ε, και το νέο της, των νέων ρυθμίσεων περί ασύλου, που τα και τα δύο έχουν μπλοκάρει στο Κοινοβούλιο. Ο ρόλος των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών είναι επίσης πολύ σημαντικός όσον αφορά τη χρηματοδότηση με την ιδέα ανάπτυξης πραγματικών εταιρικών σχέσεων για την οικονομία αλλά και για μέτρα οργανωτικά. Τώρα λοιπόν με χαρά θα ακούσουμε τα απορίσματα του φόρουμου που μπορεί να θεωρηθεί ως άμεση διαβούλευση ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών, τις ε, ε, περιφερειακές αρχές, τοπική αυτοδίκηση και τις παγκόσμιες ε, αρχές. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Νικολέτη από το EuroCities για πέντε λεπτά. Έχετε, στην κυρία Νικολέτη, με συγχωρείτε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για την πρόσκληση να σας παρουσιάσουμε τα πορίσματα της τελευταίας εκδοχής, ε, έκδοσης μάλλον του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την μετανάστευση. Ονομάζομαι Ρωσέλα Νικολέτη και είμαι υπεύθυνη συντονισμού στο EuroCities που είναι το δίκτυο των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πόλεων. Πριν να σας παρουσιάσω τα πορίσματα της έκθεσης, ε, της τελευταίας ε, έκθεσης, του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Μετανάστευσης, θα ήθελα σύντομα να σας παρουσιάσω την κύρια δομή και τους στόχους του φόρουμ αυτού. Όσους ε, κάποιοι θα γνωρίζετε ίσως ότι η πρώτη, το πρώτο φόρουμ οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2015 σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρόκειται για τη συνέχιση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ ολοκλήρωσης που γινόταν ετησίω από το 2009 μέχρι και το 2014. Το Ευρωπαϊκό Φόρο Μετανάστευσης είναι μια πλατφόρμα που μας επιτρέπει το διάλογο ανάμεσα στην, Ευρωπα... στην κοινωνία των πολιτών και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τα θέματα που αφορούν τη μετανάστευση, το άσυλο και την, την ένταξη των ε, υπηκόων τρίτων χωρών. Έχουμε λοιπόν μια φορά το χρόνο εκπροσώπους κοινωνία... της κοινωνίας των πολιτών, εκπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών αρχών και βεβαίως εκπροσώπους των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμών. Έχει αποδειχθεί σημαντική ευκαιρία ώστε οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο να παρουσιάσουν τις θέσεις τους και να τονίσουν προκλήσεις δυνατότητες βελτίωσης σε σχέση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τα θέματα της μετανάστευσης. Ο γενικός στόχος αυτού του φόρουμ είναι να βελτιώσει το συντονισμό και τη συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες ε, ε, στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι. Είπα ήδη ότι θέλει να διευκολύνει το διάλογο και ε, να παρέχει πληροφορίες για τις τελευταίες εξελίξεις της πολιτικές, επίσης να λαμβάνει στοιχεία και ε, feedback για το πώς εφαρμόζονται οι πολιτικές αυτές στην, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και να ε, δώσουν λαβές και προτάσεις για τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Επίσης, εξετάζουμε το τα στάνταρ τα οποία ε, ισχύουν επί τόπου και ε, βοηθά στο να εντοπίζονται καλύτερα ε, σχετικοί οργανισμοί, κοινωνικοί εταίροι και οι ευρωπαϊκές μας πόλεις στις προσπάθειες αντιμετώπισης των αναγκών των μεταναστών. Αυτό το φόρουμ ορίζεται, έχει μια γραμματεία και προβλέπει Έχουμε μάλλον ε, γραμματεία η οποία αποτελείται από την ε, υπαλλήλους ε, της Οικονομικής και κοινωνική επιτροπή. Έχουμε και εκλεγμένα μέλη, μεταξύ των οποίων έχω την τιμή να είμαι και εγώ. Είναι το, έτσι εξασφαλίζεται το δημοκρατικό στοιχείο στον οργανισμό και την δομή του φόρουμου που ε, πρέπει να οργανώνει τις εργασίες του ίδιου του φόρουμ και να ορίζει και την ατζέντα. Το Προεδρείο αποτελείται από έξι μέλη ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Αγγέλα, η Αγγέλα Χριστέα, ένα μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και Στη συνέχεια έχουμε και δύο εκπροσώπους της οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εμένα που εκπροσωπώ το EuroCities και το συνάδελφο από το Unity που είναι το New European Business Confederation. Έχουμε επίσης τον Φερνάντο Μπιαγκέ από το επίπεδο το εθνικό, που εξελέγει το Μάρτιο φέτος μαζί με μένα και έχουμε και την Μαρή Ντομινίκη Γεσάν που εξελέγει φέτος από την Ιταλία από την ε, Πολυπολιτισμική Ένωση Universo. Τα μέλη του Διοικητικού ε, Συμβουλίου ορίζονται για δύο χρόνια, Κλέγονται μάλλον για δύο χρόνια και δεν εκπροσωπούμε εκεί τα συμφέροντα του οργανισμού μας, αλλά ενεργούμε προς το συμφέρον του φόρουμ. Αυτά και σας ευχαριστώ και δίνω το λόγο στους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Να ακούσουμε καταρχάς από τους ε, διαφόρους καλεσμένους. Ο κ. να μας μιλήσει καταρχάς. Έχετε πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας πω ότι είναι σημαντικό αυτό το φόρουμ. Έχουμε δύσκολους καιρούς. Πολλές οι προκλήσεις. Δεν θα είναι εύκολο να μιλήσουμε για τα θέματα της μετανάστευσης. Εγώ εκπροσωπώ ε, την UNITE, μια ΜΚΟ που αγωνίζεται για την ενσωμάτωση των μεταναστών. Θεωρώ ότι ήταν ε, πάρα πολύ ενδιαφέρον το φόρουμ, γιατί για πρώτη φορά από τότε που συστήθηκε, το 2009 δηλαδή, έχει ήδη καταρτήσει 10 συστάσεις. Θα προσπαθήσω να σας τις μεταφέρω και Ελπίζω να έχουμε μια καλή συζήτηση με την Επιτροπή σας. Αποστέλλονται επίσημα αυτές οι συστάσεις ως συμβολής και των πολιτών για το μελλοντικό στρατηγικό θεματολόγιο για τη μετανάστευση. Σύντομα, να σας εξηγήσω πώς έχει διαδικασία. Ακόμη και το θέμα του φόρουμ έχει επιλεγεί μετά από δημοκρατική διαβούλευση μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Για την ε, κατάρτιση και την επιλογή των συστάσεων υπήρξαν πέντε παράλληλα εργαστήρια που συναντήθηκαν δύο φορές το καθένα και επέλεξε το καθένα δύο συστάσεις ανά ημέρα, γιατί ήταν διήμερο αυτό το, ε, αυτή η συνάντηση. Ο ρόλος των τοπικών αρχών στη διαχείριση μετανάστευσης ήταν ε, το πρώτο. Το μέλλον της μελλοντική ε, πολιτικής μετανάστευσης, δεύτερο, τρίτον, ρόλος κοινωνίας των πολιτών για την ανάπτυξη ασφαλών διάβλων, για την προστασία των μεταναστών και μια ανθρώπινη μετανάστευση, ο ρόλος τοπικών ε, κοινωνιών για τη διαχείριση μετανάστευση με χώρε εκτό Ένωση και το πέμπτο ήταν η χειραφέτηση των ε, μεταναστών για καλύτερε πολιτικέ μεταναστευτικέ. Αυτά ήταν τα θέματα. Θα σα δώσω την ιδέα του πώ συζητήθηκαν αυτά τα θέματα. Χρειάζεται αλλαγή παραδείγματο, αλλαγή σελίδα. Ποιο είναι το κόστος της μη μετανάστευσης και της μη ένταξης. Η μετανάστευση δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένα πρόβλημα προς επίλυση αλλά ως δυνητική λύση σε πολλές προκλήσεις. Ποιες είναι οι δέκα συστάσεις. Η γενική ιδέα ήταν μην λειτουργείτε ως νησίδες, ως θύλακες κλειστοί, προσπαθήστε να έχετε μία συνολική πολιτική, ε, inclusivity θα έλεγα, δηλαδή όλοι να συμπεριλαμβάνονται. Αυτό ήταν το βασικό στοιχείο που προέκυψε. Πρώτο εργαστήριο από την Παγκόσμια Τοπική Διακυβέρνηση επανάστευσε ο ρόλο των τοπικών ε, αρχών για τη διαχείριση μετανάστευσης. Πρώτη σύσταση. Να υπάρχει ρήτρα κοινωνική συνοχή στα εθνικά ταμεία για τους μετανάστες Και υποχρεωτικά ε, να συμμετέχει όλη η κοινωνία. Αυτό θα πει κοινωνική συνοχή. Ένταξη στις πολιτικές της κοινωνικής συνοχής. Δεύτερη σύσταση. Ανάπτυξη θεσμοθετημένων πλατφορμών με πολλούς ενδιαφερομένους σε τοπικό επίπεδο. Με τις τοπικές αρχές, τις ΜΚΟ, τις οργανώσεις των μεταναστών και με στόχο την παροχή αλληλέγγυων υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του καθεστώτος. Σαφές το μήνυμα και εδώ τοπικό οικοσύστημα υποστηρικτικό αλληλέγγυο και πάλι όχι θύλακες, όχι νησίδες απομονωμένες, αλλά συντονισμένη δράση. Αυτό είναι το σαφές μήνυμα της δεύτερης σύστασης. Τρίτη σύσταση. Από το δεύτερο εργαστήριο, το μέλλον δηλαδή ε, της μελλοντικής πολιτικής της Ένωσης για την νόμιμη μετανάστευση. Δομημένη διαδικασία για τη διαβούλευση με τοπικές αρχές ΜΚΟ και κοινωνικούς εταίρους για τη διαχείριση της νόμιμη μετανάστευση. Τέταρτη σύσταση. Να προσαρμοστεί η οριζόντια οδηγία με εναρμόνιση των όρων υποδοχής και ε, για όλους τους ε, ε, μετανάστες ανεξαρτήτως του κράτους από το οποίο προέρχονται. Επίσης, κινητικότητα, να υπόψη και οικογενειακή επανένωση. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάλι υπάρχουν απομονωμένοι θύλακες και εμείς θα θέλαμε να υπάρξει μια εναρμόνιση. Αυτό λέει η κοινωνία των πολιτών στο, στην τέταρτη σύσταση, της πέμπτη σύσταση, από το τρίτο εργαστήριο, το ρόλο των γνώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την ανάπτυξη σαφών διάβλων, για λόγους προστασίας και ανθρώπινης ε, συμπεριφοράς και μετανάστευσης. Τα προγράμματα της Γενικής Επανέλευσης πρέπει να είναι συμπληρωματική δρόμη για την προστασία. Το έκτο, έκτη σύσταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να πάρει μέτρα για την εναρμόνιση των διαδικασιών των κρατών μελών, για την υποδοχή και την ένταξη των μεταναστών ανεξαρτήτως του πώς έφτασαν και από πού προέρχονται. Για να δοθούν επίσης, ε, ε, να δοθεί θέση προσοχή στις ευάλωτες ομάδες και να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η χρηματοδότηση του νέου πιδελταπή για τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας, καθώς και των τοπικών αρχών. Έβδομη σύσταση από το τέταρτο εργαστήριο, ρόλος κοινωνίας των πολιτών και άλλων μη δημόσιων φορέων για τη βελτίωση της συνεργασίας με χώρες εκτός Ένωσης για τη διαχείρισή της μετανάστευση, ενίσχυση με οργανώσεις της διασπόρας και της κοινωνίας των πολιτών, υποστήριξη των προσπαθειών τους για την παροχή πληροφόρησης και κινήτρων για την επανένταξη των μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους. Εδώ το μήνυμα είναι να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί μια μεταναστευτική πολιτική και για τους μετανάστες αλλά και μαζί με τους μετανάστες. Όγδοη σύσταση. Να προωθηθεί ο περιφερειακός διάλογος και πλατφόρμες για να δημιουργηθούν ΣΔΙΤ για την κινητικότητα, συμπράξεις δημοσιοδοτικού τομέα δηλαδή. Και τελευταίες δύο στάσεις από το πέμπτο εργαστήριο για την χειραφέτηση των μεταναστών, για καλύτερε και πιο ορκωμένε πολιτικέ μετανάστευση. Πιλωτικά προγράμματα πρέπει να εφαρμοστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλε τι περιφέρειε, ώστε πρόσβαση στα δικαιώματα να είναι γενική. Και να βοηθήσουν και οι μετανάστες την κοινωνική. Και τέλος, να στηριχθούν οι τοπικές κοινωνικές ε, οργανώσεις, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών για να προωθηθούν πολιτικές και δράσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου στο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με την πολυτομιακή και πολυπαραγοντική προσέγγιση. Ε, ήσασταν λίγο πιο ε, στην παρέμβασή σας, ξεπεράσετε τα πέντε λεπτά, αλλά τέλος πάντων. Ήταν σημαντικό που ακούσαμε όλες τις συστάσεις του φόρουμ και νομίζω θα βοηθήσει αυτό και στη συζήτησή μας Σα Ευχαριστώ. Άρα μην ανησυχείτε που ξεπέρασε το χρόνο. τελευταίο ο μιλητής, Πουρβουλέσκου, από την ΕΟΚΕ. Πέντε λεπτά. Σα ευχαριστώ πολύ. Προτιμώ να μιλήσω στα γαλλικά. Εάν δεν κατανοείτε τα γαλλικά, παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας. Κυρία Πρόεδρε, Αγαπητοί τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΠΕ, είμαι πολύ ευτυχής που μπορώ να σας μιλήσω για αυτό το φόρουμ της μετανάστευσης, όπως η συνάδελφος ήδη σας εξήγησε. Ξεκινήσαμε τη δουλειά αυτή όσον αφορά τη διαβούλευση της κοινωνίας των πολιτών πριν από 11 χρόνια το 2009 όπου οργανώσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πρώτο φόρουμ της μετανάστευσης ανάμεσα το 2009 και το 2014 και τότε το, πολύ πριν από την ε, μεταναστευτική κρίση αρχίσαμε να ασχολούμαστε με τη μετανάστευση. Η ιδέα μας ήταν να έχουμε μια συνεργασία με τις οργανώσεις της που εργάζονται για αυτά τα θέματα. Γιατί όσον αφορά την τεχνική πτυχή, συζητήσαμε και εγκρίναμε σχετικές νομοδοτήσεις από τη δεκαετία του 80 αλλά ανέκαθεν θεωρούσαμε πως είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να οργανώσουμε ε, δημόσιες ακροάσεις με τα ευρωπαϊκά δίκτυα, αλλά και να οργανώνουμε, ε, να οργανώσουμε μάλλον μια ευρωπαϊκή συζήτηση. Γι' αυτό και προτείναμε στην Κομισιόν από το 2008 να διοργανώνεται ετησίως αυτή η συνεδρίαση. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία ώστε να έχουμε την αντίδραση της κοινωνίας των πολιτών και κάθε χρόνο συζητάμε για πολύ σημαντικά θέματα. Πάντοτε έχουμε κάνει προτάσεις στην Επιτροπή. Έχουμε πάντοτε μία εικόνα πιο ε, συγκεκριμένη και πιο λεπτομερή όσον αφορά την μετανάστευση, αλλά έχουμε παρατηρήσει ε, ότι οι λαϊκιστές είναι αυτοί που κερδίζουν πάντα και γι' αυτό είναι σημαντικό να ακούμε την κοινωνία των πολιτών και τις συστάσεις του φόρουμ Διοργανώνουμε το χρόνου το φόρουμ τον Ιούνιο και ελπίζω ότι η ΛΥΜΠΕ και το Κοινοβούλιο θα συμμετέχουν ε, δραστήρια γιατί πέρσι ήταν οι ευρωεκλογές, ε, ήταν η αλλαγή της Κομισιόν και δεν πήγε πολύ καλά ε, το πράγμα. Ελπίζω όμως πως θα μπορέσουμε μαζί να προτείνουμε κάτι πιο συνεκτικό όσον αφορά την μετανάστευση. Γιατί βλέπουμε ακόμα και στην ΟΚΕ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αντιδράσεις ε, εχθρικές στην μετανάστευση. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η μετανάστευση είναι εξαιρετικός πόρος, πλούτος για την Ευρώπη, πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά ότι η μετανάστευση δεν είναι ενάντια καθόλου στο ευρωπαϊκό όραμα και γι' αυτό ελπίζω πως ακόμα και η νέα Επιτροπή θα εργαστεί μαζί μας, θα συνεργαστεί μαζί μας, ώστε να υλοποιηθεί το επόμενο φόρουμ. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ε, ποιο θα είναι το πρόγραμμα γιατί θα πρέπει όλα αυτά να διοργανωθούν με τη συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Έχουμε φυσικά προτάσεις, αλλά από κοινού θα ορίσουμε τα θέματα για τον επόμενο χρόνο. Επίσης θα αλλάξουμε εταίρο στην Κομισιόν, είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο δηλαδή, αλλά ελπίζω ότι το φόρουμ θα διοργανωθεί πολύ καλά. Γι' αυτό προτείναμε τον Ιούνιο και όχι τον Απρίλιο όπως ε, συνηθίζαμε, γιατί από το 2015 το φόρουμ οργανωνόταν τον Απρίλιο. Θεωρώ πως αυτός ο τρόπος είναι ένας τρόπος με εξαιρετικά δυναμικό για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ελπίζω πως η συζήτηση τώρα θα διευρύνει την εικόνα που έχουμε για τα θέματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν, ειδικά δεδομένων των άλλων συζητήσεων που είχαμε σήμερα το πρωί. Ε, πολύ έντονες ε, συζητήσεις, καμιά φορά ξεχνάμε τα βασικά τα οποία αναφέρατε. Ε, θα τα πω με δικά μου λόγια. Ε, πρώτα απ' όλα η μετανάστευση είναι κάτι το οποίο πάντα υπήρχε και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι Ευρωπαίοι πολίτες πάντα πηγαίνουν σε άλλα μέρη του κόσμου για να φτιάξουν τη ζωή τους. Οπότε ίσως η πραγματική πρόκληση δεν είναι ο αριθμός των προσφύγων αλλά πώς να το διαχειριστούμε και σαφώς είπατε στην εισαγωγή σας ότι ε, για να γίνει μια σωστή διαχείριση απαιτούνται όλοι. Το εθνικό επίπεδο, το τοπικό επίπεδο, οι αρχές, ε, ΜΚΟ, τα άτομα και οι πολίτες ε, και οι πρόσφυγες για να το οργανώσουν και να διασφαλίσουμε την ένταξη αυτών που θα μείνουν για να ωφεληθούμε όλοι και ως ε, Γερμανίδα γνωρίζω ότι στον παλιό τηλεφωνικό κατάλογο βλέπουμε διάφορα ονόματα που λέμε ναι είναι Γερμανός αυτός αλλά ίσως να έχει έρθει η Γερμανία πριν από δεκαετίες. Ας κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε και η εμπειρία από το μέτωπο θα έλεγα είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε γιατί γνωρίζετε και τις προκλήσεις ε, και τις ε, λύσεις και ίσως συχνά δεν εστιάζουμε στην ε, εμπειρία στο, στο μέτωπο θα έλεγα στις κοινότητες. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για την παρουσίασή σας. Κοιτάω τώρα εδώ γύρω Δεν ξέρω τώρα αν σας αρκούν τα ευρήματα. Ή αν έχετε κάποια ερώτηση. Αλλιώς θα κάνω εγώ. Με όλη τη δουλειά που έχετε κάνει, σε εργαστήρια, σε συναντήσεις, έχοντας κατά νου το ότι η Κομισιόν προσφέρει, ετοιμάζει αυτό το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση, θα πρέπει να βρούμε τρόπο διαχείρισης της εισερχόμενης ε, μετανάστευσης ε, ε, και των ετούντων άσυλο και να βελτιωθεί και η νόμιμη μετανάστευση και απασχόληση. Οπότε η πρώτη μου ερώτηση είναι ε, έχετε κάποια επαφή με την παλιά κομισιόν, ε, την νέα κομισιόν ε? δεν ξέρω αν έχετε κάποιες ιδέες, συμβουλές που θέλετε να δώσετε στην κομισιόν. Ίσως πριν ή μετά όπως προτιμάτε. Ε, αν είναι... Δεν ξέρω, θέλετε να προσθέσετε κάτι ή πριν ή μετά. Όχι. Όχι για την ώρα. Οπότε θα ακούσουν τις συμβουλές που θα δώσετε εσείς, εάν θέλετε να δώσετε κάποια περαιτέρω πληροφορία. Εγώ μπορώ να πω ότι το φόρουμ είναι μια πάρα πολύ καλή ε, βάση για ανταλλαγή πληροφοριών και ως εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών ε, θεωρούμε ότι η Κομισιόν και η Επιτροπή ε, μας ακούνε Και νομίζω ότι η έκθεση αυτή μπορεί να αποτελέσει μια καλή βάση για να ξεκινήσει ένας διάλογος για να συζητήσουμε ακριβώ και τα μελλοντικά στοιχεία ενός μελλοντικού συμφώνου για τη μετανάστευση. Υπάρχουν ε, κάποια σημεία που ξεκάθαρα έδειξαν ότι μπορούν να έχουν μεγάλη σημασία και υπάρχει μια ανάγκη εναρμόνισης θα έλεγα και η ανάγκη να μην εργαζόμαστε απομονωμένοι αλλά να έχουμε μια συνολική προσέγγιση στα θέματα αυτά περιλαμβανωμένη του συντονισμού, της συνεργασίας μεταξύ κοινωνίας των πολιτών, των πόλεων, των περιφερειών, των κοινωνικών εταίρων, ΜΚΟ και των πολιτών. Οι πολίτες ε, τα ζητάνε αυτά. Θέλουν να υπάρχει το θέμα αυτό της ένταξης ε, να περιληφθεί σε μια ευρύτερη συζήτηση για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική συνοχή. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι γεγονός ότι η Κομισιόν στηρίζει και συνδιοργανώνει το φόρουμ, οπότε ε, παρά το ότι θα έπρεπε να είναι προφανές και εγώ το κατάλαβα, θα ήθελα να ρωτήσω στην Κομισιόν αν μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι βεβαίως το φόρουμ αυτό θα είναι στην ημερήσια διάταξη για το μελλοντικό έργο της νέας Κομισιόν. και να δούμε βεβαίω ε, το τι σκοπεύει να κάνει και η Κομισιόν στην επόμενη φάση. Καλησπέρα σα. Βενσόν Κατό λέγομαι, οργάζομαι στην ομάδα ένταξης ε, της γενική διεύθυνση Εσωτερικών. Σας ευχαριστώ που οργανώσετε αυτήν την συζήτηση. Όπως είπαν και οι ομιλητές, ε, υπάρχει δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Κομισιόν να διοργανώνεται αυτή η ετήσια εκδήλωση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Εδώ και χρόνια οργανώνουμε από κοινού αυτή την εκδήλωση. Εκατοντάδες οργανώσεις ε, έχουν λάβει μέρος. Εγώ ήμουν ε, στην ομάδα που διοργάνωσε το πέμπτο φόρουμ υπήρχε αυτό το φόρουμ ακριβώς για την συζήτηση, όχι μόνο οργανώσεων ε, που μπορούσαν να μιλήσουν με την Κομισιόν, αλλά και η Κομισιόν ε, και οι άλλοι. Ε, είναι μέρος της συζήτησης. επίση ε, αυτά τα έχει τονίσει και η κυρία Φόντερ Λάιεν ε, και η Επιτροπή Αρμόδη με έχουν μιλήσει για ένταξη που είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Νέας Κομισιόν. Επίσης θα έλεγα ότι λαμβάνουμε υπόψη ε, την συζήτηση αυτήν ως μια συνεχή διαδικασία Έχουμε διάφορα θέματα. Το τέταρτο φόρουμ, παραδείγματο χάρη, εστίασε στην ένταξη στην αγορά εργασία. Έχουμε λοιπόν αυτή την ατζέντα και θα χρησιμοποιήσουμε και αυτές τις συστάσεις για να σκεφτούμε τα μελλοντικά βήματα. τώρα οργανώνουμε το έκτο φόρουμ. Ενθαρρύνουμε λοιπόν τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών να έρθουν να μας ενημερώσουν για τις προτάσεις αυτές, τα προτινόμενα θέματα. Τα προτινόμενα θέματα βασίζονται σε μια συζήτηση που έλαβε χώρα στο πέμπτο φόρουμ και σε μια έρευνα που κάναμε με τα μέλη του πέμπτου φόρουμ. Για να δούμε τι θα έπρεπε να συζητήσουμε. Και στο πλαίσιο αυτό να έχουμε προτείνει να συζητήσουμε τις πτυχές κοινωνικής ένταξης ως μια πιο γενική προσέγγιση. Επίσης αναφέρουμε τις ε, νόμιμες ε, διόδους ε, και Σας Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ για την παρέμβασή σας αυτή. Ε, θέλει να μιλήσει και ο συνάδελφος εδώ βλέπω. Ευχαριστώ. Είμαι νέος βουλευτής, συγγνώμη. Και πάω από τη μια συναντρία στην άλλη, τρέχοντας. Γι' αυτό δεν ήμουν ε, και από την αρχή εδώ. Χαίρομαι πάντως ε, που οι συλλογικότητε έχουν τη θέση τους εδώ για 18 χρόνια. Ήμουν στη Βόρεια Γαλλία, 30 χιλιόμετρα από το Καλέ, δήμαρχος και πριν έρθουν οι Σύριοι πρόσφυγες το 2015, γιατί δεν μπορούσε τότε το κράτος να αντιδράσει με τους ε, γιατρούς χωρίς σύνορα. Αυτά τα 2.500 άτομα, μέσα σε 23.000 που είμαστε, δημιουργήσαμε αυτόν τον καταβλισμό. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη οι συλλογικότητες για τις αποφάσεις και πράγματι έχουν να αντιμετωπίσουν οι αιρετοί ε, πολλές δυσκολίες για τη διαχείριση των ατόμων που φτάνουν στην επικράτειά τους. Ο Δήμαρχος ουσιαστικά είναι στην πρώτη γραμμή. Ήμουν ε, στη Σάμο ε, πριν τρεις εβδομάδες. Ο Κακομύρης, ο Δήμαρχος, ε, τον έχει ξεπεράσει η κατάσταση και είναι και το μαξιλάρι ανάμεσα στον πληθυσμό και τους μετανάστες. Πρέπει λοιπόν να τα δούμε αυτά ε, και να έχουμε μια ευαισθησία απέναντι στι λογικότητε. Όταν τα κράτη-μέλη κάποια στιγμή, δυστυχώ δεν είναι παρόντα, έστω να βοηθήσουμε τι λογικότητε. Εγώ αναζητούσα χρηματοδότηση γιατί 4,5 εκατομμύρια έκανα αυτού του κατάχρησμού που έφτιαξα και σε μεγάλο βαθμό χρηματοδοτήθηκε από τα ταμεία του Δήμου. Βοήθησαν οικονομικά και γιατροί χωρί σύνορα. Δεν είναι λογικό αυτό όμω, γιατί δεν είναι δική μα αρμοδιότητα. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε καμιά χρηματοδότηση τότε από την Ευρώπη. Πραγματικά είμαι πολύ, έτσι, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα ε, και έχω ιδιαίτερη ευαισθησία. Για την ένταξη αυτών των ανθρώπων πρέπει να παίξει το ρόλο τους ε, τα κράτη και οι συλλογικότητε και οι ΜΚΟ και οι ενώσεις. Ο πληθυσμό. στη Γαλλία δημιούργησα την Εθνική ε, Ένωση των Εδαφών που φιλοξενούν ε, για να προωθήσουμε ακριβώς την υποδοχή, γιατί είναι πλούτος αυτό που έχουν να μας προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι σημαντικό. Και κάτι άλλο στο οποίο επιμένω. Για να μας βοηθήσετε, πρέπει να έχουμε και το σωστό αφήγημα, τη σωστή γλώσσα. Μην δημιουργούμε φόβο Μπορούμε να δημιουργήσουμε αποδοχή μόνο και μόνο με τις λέξεις. Αν μιλάμε για πλημμύρα και ρεύματα μεταναστευτικά, πανικοβάλλονται όλοι. Αν λέμε όμως πρέπει να υποδοχθούμε 200 200-300 χιλιάδες ή ένα εκατομμύριο, όταν είμαστε 500 εκατομμύρια δεν και πια και τόσο τραγικό, μπορούμε να το κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το φόρουμ των τοπικών αρχών. ήμουν στο πέμπτο, ελπίζω να είμαι στο έκτο. Και θα έρθω να σας δω. Έχουμε και το Παγκόσμιο Φόρουμ σε 15 μέρες. Και εκεί ζήτησα να δω αν υπάρχει θέση για τις λογικότητες και με διαβεβαίωσαν ότι θα συζητηθεί στη Γενέβη. Τουλάχιστον εγώ θα επαγρυπνώ. Και θα βλέπω τι αποφάσεις λαμβάνονται ώστε να είναι παρούσες και συλλογικότητες. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Δεν ήταν και ερώτηση αυτό βέβαια, αλλά ήταν μια πολύ καλή προσθήκη στα όσα συζητήθηκαν στο φόρουμ. Και συμφωνώ απολύτως ότι οι κοινωνίες οι τοπικές, οι δήμοι και οι κοινότητες έχουν πολύ σημαντικό ρόλο και το λέω και από τη, από τη γερμανική σκοπιά. Χωρίς ΜΚΟ και χωρίς τοπική κοινωνία το πρόβλημα θα ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αντιμετωπίσαμε το 2015 και τα επόμενα χρόνια. Και Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο στηρίζει ακριβώς αυτή την άποψη. Οι τοπικές κοινωνίες δηλαδή είναι σημαντικές και πρέπει να υποστηριχθούν και οικονομικά με προπολογισμό. Δεν είναι τα πάντα το χρήμα, καλό είναι και αυτό και χρειάζεται, αλλά και η διευκόλυνση των διαδικασιών και η κάλυψη όλων των προποθέσεων ε, για το κατάλημα, για την ένταξη κτλ. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν σε όλα τα επίπεδα. Θέλετε εσείς κάτι να προσθέσετε ή αυτό ακριβώς συζητήθηκε στο φόρουμ. Μάλιστα. Προφανώς έτσι έγινε. Άρα, περιμένουμε με αρπομονησία το επόμενο φόρουμ. Και θα σας ξανακαλέσουμε είτε εσάς τους ίδιους είτε άλλους εκπροσώπους θα δούμε. Ελπίζουμε να αλλάξει η κατάσταση τα επόμενα χρόνια και να έχουμε και κάποιες άλλε ιδέες στο μεταξύ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ φέτο εσείς. Καλή τύχη για το επόμενο φόρουμ. Να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση τοπική κοινωνία. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Um, colleagues, the next point of our agenda... Συνάδελφοι, το επόμενο σημείο της σημερινής μας διάταξης θα ξεκινήσει στις 3.45. Οπότε τώρα έχετε λίγο καιρό για να πάρετε αέρα έξω. Αλλά να θυμάστε ότι δεν είναι το τέλος της σημερινής μας συνεδρίασης, οπότε σας παρακαλώ στις 3.45 να είστε εδώ για το επόμενο σημείο στην ημερήσια μας διάταξη. Mm-hmm. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Allora, colleghi, cari colleghi, buon pomeriggio. Λοιπόν, καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι για το θέμα αυτό αντικαθιστώ τον πρόεδρο, τον Λόπες Αγγιλάρ, οπότε έχω την χαρά να διευθύνω την συζήτηση. Περνάμε λοιπόν σημείο 9, το οποίο αφορά ανακοίνωση από την Κομισιόν για τις ε, διατάξεις προστασίας προσωπικών ε, δεδομένων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έναν απολογισμό. Πρόκειται για μια διαδικασία στο πλαίσιο του GDPR του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Το άρθρο 97 προβλέπει ότι η Κομισιόν κάνει μια πρώτη αξιολόγηση του σχετικού κανονισμού ε, το 2020 και υποβάλλει αυτήν την αξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε εδώ πέρα έχουμε τον κύριο Λιβιέρ Μικόλ και τον Μπρούνο Τζακαρέλη της ε, Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, ο οποίος καλώς ορίζω, οι οποίοι θα παρουσιάσουν αυτήν την ανακοίνωση. Οπότε θα δώσω αμέσως ε, τον λόγο πρώτα στον κύριο Μικόλ εδώ πέρα για να μας ε, κάνει μια εισαγωγή στην συζήτηση. Έχετε τον λόγο. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω την ανακοίνωση και τη δουλειά μας ε, που σχετίζεται με την ε, αξιολόγηση του άρθρου 97 του κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η ανακοίνωση που δημοσιεύσαμε τον Ιούλιο είναι κομμάτι της αυστηρής παρακολούθησης του κανονισμού που κάνει η Κομισιόν. Το σκεπτικό λοιπόν ήταν να γίνει μια ανασκόψη της εφαρμογής από τα κράτη-μέλη. και να προετοιμαστούμε για την αξιολόγηση που θα εκδοθεί το 2020. Οπότε αυτό δείχνει τη σημασία που αποδίδει η Κομισιόν σωστή εφαρμογή του κανονισμού αυτού. Πρώτα απ' όλα είχα μια σειρά διμερών διαλόγων με τις εθνικές αρχές για την εφαρμογή της εθνικής ε, νομοθεσίας. Και βεβαίως έχουμε τον διάλογο που περιλαμβάνει και την κοινωνία των πολιτών. Επίση υπάρχει το θέμα του Ευρωβαρόμετρου, το οποίο ερευνά ακριβώ το κατά πόσο γνωρίζουν οι πολίτε τον σχετικό κανονισμό. Πού βρισκόμαστε λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα. Ένα κράτος μέλος ακόμα δεν έχει περάσει εθνική νομοθεσία. Από την άλλη, ο κανονισμός έχει επεκταθεί και στις χώρες ΕΖΕΣ μετά από μια συμφωνία που περιλαμβάνει τις χώρες ΕΖΕΣ ε, βλέπουμε ότι το νέο σύστημα διακυβέρνησης ε, έχει αρχίσει να αποδίδει. Είναι μια διαδικασία βεβαίως που χρειάζεται χρόνο, αλλά βλέπουμε ότι οι αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων τα παίρνουν τα πράγματα στα σοβαρά ξεκινάνε τώρα να χρησιμοποιούν τις νέες τους αρμοδιότητες και σταδιακά χρησιμοποιείται αυτός ο μηχανισμός. Βεβαίως, ε, η βασική απόφαση που θα πρέπει να λάβουν αυτές οι αρχές ε, είναι κάτι το οποίο ακόμα ερευνούν και αναμένουμε ότι τόσο σημαντική απόφαση θα ληφθεί προς το τέλος του έτους ή αρχές του επομένου. Κάτι το οποίο είναι επίσης σημαντικό είναι να δούμε το ότι ε, οι πολίτες ε, χρησιμοποιούν περισσότερο και ασκούν τα δικαιώματά τους. Ζητάμε, παραδείγματος χάρη, να ζητούν πρόσβαση στα δεδομένα τους ε, ή έχουμε δει Μίκιο οι οργανώσεις ε, καταναλωτών να χρησιμοποιούν την δυνατότητα να ε, έχουν παραδείγματο χάρη ε, εκπροσώπηση κατά τέτοιων εταιριών, κατά το οποίο ξεκίνησε αμέσως και συνεχίζεται ακόμα και μπορεί να δούμε και ακόμα περισσότερα εάν περάσει η οδηγία περί αντιπροσωπευτικής ε, δράσης. Γιατί έτσι θα γίνει ακόμα πιο εύκολο για ΜΚΟ να αναλαμβάνουμε έτσι συλλογική δράση. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, πολλές από τις ανησυχίες ε, που είχαν εκφραστεί πριν ε, τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός τελικά δεν υλοποιήθηκαν. Είδαμε κάποιες εταιρείες οι οποίες ε, λένε ότι είναι αυτό ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους ε, ανταγωνιστές τους. Και βεβαίως ε, γνωρίζουμε την ανησυχία μικρών και μεσαίων εταιριών και κάτι το βασικό είναι το ότι θα πρέπει να τους στηρίξουμε με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Έχουμε ακριβώς ε, αυτά τα εργαλεία που δίνουν οι αρχές ε, προστασίας προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει ένας κώδικας συμπεριφοράς, μπορεί να βοηθήσει για να στηρίξουμε την συμμόρφωση με τον κανονισμό υπόδειγμα ε, ρήτρα ε, στις συμβάσεις, επίσης ε, πράγματα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να στηρίξουμε την εφαρμογή, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό δεδομένης της αξιολόγηση είναι το ότι η προστασία δεδομένων είναι αναπόσπαστο μέρος διαφόρων πολιτικών στον τομέα της υγείας όπου έχουμε ευαίσθητα δεδομένα όταν μιλάμε για ηλεκτρονικά αρχεία υγείας στον τομέα της μεταφοράς, με τα συνδεμένα αυτοκίνητα, της ενέργειας, με τους έξυπνους μετρητές. Ε, το βασικό είναι οι αρχές αυτές να ενσωματώνονται σωστά στην τομεακή πολιτική. Οπότε τώρα εξετάζουμε την αξιολόγηση το 2020 το μήνυμα που έχουμε αυτήν την ε, στιγμή είναι το ότι ακριβώς ε, έχουμε το θέμα του κανονισμού αυτού μια στιγμή της επιβολής ε, δεν είναι η στιγμή για να αλλάξουν δραστικά οι κανόνες αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είμαστε πιο συνεπείς στην εφαρμογή και αυτό πράγματι θα κάνουμε. Θα έχουμε και την συνεισφορά του Συμβουλίου στις αρχές του επόμενου έτους και βεβαίως ε, θα συμβουλευτούμε και τους ενδιαφερόμενους. Και βεβαίως ε, με αυτό αναμένουμε και τις απόψεις του Κοινοβουλίου Θα ήθελα τώρα να στραφώ στον Μπρούνο για τη διεθνή διάσταση και την εξαγωγή του μοντέλου μας σε άλλες χώρες. Ναι. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ Δόκτωρ Μίκολα και θα δώσω το, λόγο στον κύριο Τζιγκαρέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσουμε σύντομα να μιλήσουμε για τη διεθνή πτυχή, για διάσταση μάλλον, ε, το τι μπορούμε να αποκομίσουμε δηλαδή από διεθνούς απόψεως ε, για την εφαρμογή του GDPR και μετά θα δούμε ποιες είναι οι θετικές αξιολογήσεις ε, που έχουμε πάρει για να δούμε ποιες θα είναι οι θετικές εξελίξεις για το GDPR. Όταν μιλάμε για την ερμηνεία, ο καιρός ε, έχει αλλάξει. Ε, κάποιοι από εσά ε, θα θυμάστε ότι όταν ξεκινήσαμε αυτό το εγχείρημα, συχνά Ακούγαμε παντού, α, αυτό είναι ευρωπαϊκό θέμα, ε, η ιδιωτικότητα είναι ευρωπαϊκή έννοια. Όμως δεν ισχύει πια αυτό. Οι διάφορες χώρες στον κόσμο ολόκληρο, σε πολλού, πολλά διαφορετικά μέρη του κόσμου έχουν διαπιστώσει ότι στην ψηφιακή εποχή όλοι αντιμετωπίζουμε παρόμοιες προκλήσεις και παρόμοιες ε, ευκαιρίες. Βέβαια, ε, όλοι πρέπει να κατανοήσουμε ότι ε, τα δεδομένα πλέον θεωρούνται και ως ε, προϊόν και ε, βεβαίως η προστασία αυτών είναι επιτακτική ανάγκη γιατί ε, η κακή χρήση των στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε παραποίηση της δημοκρατίας, να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν λειτουργεί η ψηφιακή οικονομία. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία είναι πια προβλήματα για ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και βέβαια σημαίνει και νέες ευκαιρίες και για την προστασία των δεδομένων ε, των πολιτών, εφόσον τα δεδομένα κυκλοφορούν γιατί λένε και περισσότερες χώρες στον κόσμο υιοθετούν ή εξυγχρονίζουν την νομοθεσία τους και την καθιστούν παρόμοια με τη δική μας, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή στοιχείων όχι μόνο για το εμπόριο αλλά και για την συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών. Και εμεί στι Κομισιόν μαζί με τους διεθνεί μας εταίρους προσπαθώντα να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη σύγκληση επί τη βάση βασικών στοιχείων, να έχουμε δηλαδή μια γενική νομοθεσία για τα δεδομένα, δικαιώματα τα οποία είναι ε, δυνατόν να επιβληθούν, να έχουμε αρχή προστασία δεδομένων, Έχουμε λοιπόν ανακοινώσει και αναπτύξει ατζέντα από το 2017 με τον ανακοινωθέν για την προστασία των δεδομένων σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο και από αυτή τη ατζέντα δουλεύουμε έκτοτε και διερευνούμε τη δυνατότητα υιοθέτηση υιοθέτηση ε, αποφάσεων με καταλληλότητες με τέτοιες χώρες που έχουν προοδεύσει σε αυτό το τομέα και αυτό έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα η υιοθέτηση της συμφωνίας <laughs> καταλληλότητας με την Ιαπωνία, η οποία υπεγράφει φέτος ε, που δημιούργησε έτσι τον μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη περιοχή μεγα, ελεύθερης και ασφαλούς ροής δεδομένων ανάμεσα σε χώρες. Με την Κορέα, Κορέα είμαστε σε ένα αρκετά προηγμένο στάδιο και μάλλον θα ολοκληρωθούν οι συζητήσεις ε, ε, στο τέλος του χρόνου Επίση, ανταλλάσσουμε σχετικέ ε, ε, πληροφορίε με τι χώρε τη Λατινική Αμερική για σύναψη παρόμοια συμφωνία. Ε, το ίδιο με χώρε τη Ασία, όπω η Ινδία, η Ινδονησία και η Ταϊβάν, όπω και με χώρε τη νότια και ανατολική μα γειτονία, αλλά και με τι χώρε τη Αφρική, η οποία, όπω ξέρετε, ζει μια φοβερή ψηφιακή άνθηση. Ρυθμίσεις δηλαδή που διευκολύνουν πάντοτε τις ροές δεδομένων. Και όπως είπα, προς όφελος ε, έτσι ώστε να έχουμε προς όφελος λοιπόν των πολιτών αλλά και της προστασίας των δεδομένων των πολιτών. Ε, συνεργαζόμαστε με τους ενδιαφερόμενους φορείς, ε, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων για να μπορέσουμε να χειραγωγήσουμε το πλήρες δυναμικό ε, της μεταφοράς δεδομένων. Και αυτό σημαίνει και εργασία όχι μόνο για την καταλληλότητα, αλλά και για στάνταρ συμβατικές ρήτρες που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες τις καθημερινές τους δραστηριότητες, πιστοποίηση, και άλλοι μηχανισμοί για τις μεταφορές. Φυσικά θα προσέχουμε πολύ στις εκκρεμείς ε, υποθέσεις ε, και τις αποφάσεις που περιμένουμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τους ερχόμενους μήνες, ώστε να έχουμε διάφορες διευκρινήσεις για τα ακριβή στάνταρ που πρέπει να εφαρμόζουμε όταν ε, χρησιμοποιούμε τους μηχανισμούς μεταφοράς. Άλλη σημαντική πτυχή της δουλειάς μας αφορά την, ε, το συντονισμό ανάμεσα στην προστασία δεδομένων και το εμπόριο. Εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα σύστημα το οποίο έχει στόχο να εξασφαλίσει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας, ενώ ταυτόχρονα παραμένει ανοιχτό στις μεταφορές δεδομένων. Έχουμε Επίσης, ε, χειριστεί την ψηφιακή προστασία, δηλαδή δεν νομίζουμε ότι η πλήρης αποθήκευση δεδομένων έχει να κάνει με η απαγόρευση χρήση δεδομένων, έχει να κάνει με την προστασία των δεδομένων. Έχουμε λοιπόν συμφωνίες ε, Έχουμε διαπραγματεύσεις στον ΠΟΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο αποκλεί, η οποία συμφωνία αποκλεί την παράβαση των ε, δικαιωμάτων. Είμαστε αποφασισμένοι. Τα ανθρωπίνα δικαιώματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν μπορούμε να τα διαπραγματευτούμε στα μπορικά μέσα και χρειαζόμαστε και την κατάλληλη γλώσσα που να τα αναγνωρίζει όλα αυτά. Επίσης είναι χρήσιμο να χρησιμοποιηθεί αυτό το μέσο ώστε να καταπολεμηθούν μέτρα τα οποία δεν έχουν σχέση με την προστασία των δεδομένων αλλά ε, εκμεταλλεύονται την προστασία των δεδομένων για να πετύχουν άλλους ε, σκοπούς. Επίσης φαίνεται ότι έτσι υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία μπορεί να συμπληρώνουν, να, να συγγνώμη. Τέλος, ε, αυτό που κάνουμε από φέτος είναι ότι ενώ η σύγκληση γίνεται, υπάρχει, είναι πραγματικότητα, γιατί σε άλλους τομείς βλέπουμε αποκλήσεις, διαφορές, Έχουμε ένα τομέα όπου μπορούμε να δούμε αυξανόμενη σύγκληση, αυξανόμενη σύγκληση η οποία όμως ε, ε, φέρνει ε, αποτελέσματα. Υπάρχει όμως ένα κεφάλαιο που λείπει, δηλαδή είναι η συνεργασία ανάμεσα στις αρχές επιβολής. Σήμερα μεγάλες παραβιάσεις στοιχείων ή πιο βλαβερές καταχρήσεις των στοιχείων των δεδομένων επηρεάζουν πολίτες και κάποιες φορές εκατομμύρια πολιτών ταυτόχρονα σε διάφορες ε, δικαιοδοσίες. Και δεν έχει νόημα καθόλου, ας πούμε, για το Facebook και την Cambridge Analytica. Οι δικές μας, οι δικές αρχές προστασίας δεδομένων δεν συνεργάζονται περισσότερο με άλλες αρχές ε, προστασίας δεδομένων στον κόσμο που διερευνούν για να το σταματήσουν αυτό στη σωστή στιγμή. Αυτό υπάρχει σε άλλους ρυθμιστικούς τομείς, ας πούμε, στην ε, ανταγωνισμό ή στα θέματα αντιτράστα. Υπάρχουν συστήματα συνεργασίας. Είναι κάτι που αν θέλουμε να έχουμε αποτελεσματική επιβολή, το είπε και ο συνάδελφος Ολιβιέ Μικόλ, ότι δηλαδή χρειάζεται να υπάρχει αποτελεσματική επιβολή όλων αυτών εντό τη Ένωση και βεβαίως πρώτα πρέπει όλα αυτά να λειτουργήσουν καλά εδώ, όταν λοιπόν έχουμε να κάνουμε με τόσο σημαντικά θέματα ασφάλειας Αυτό σημαίνει περισσότερη αμοιβαία συνεργασία ανάμεσα στην Ένωση και τις ε, άλλες επιοπτικές αρχές. Έχουμε στο GDPR το άρθρο 50 της, ε, της ε, οδηγίας του κανονισμού, με συγχωρείτε, και όχι το άρθρο 50 της συνθήκης που είναι διάσημο για άλλους λόγους. Προβλέπετε λοιπόν ότι ε, αυτό είναι το άρθρο το οποίο, το οποίο θα μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες. Τέλος, αξιολόγηση. Ποια είναι η διεθνής πτυχή της αξιολόγησης ε, που ετοιμάζει η Κομισιόν. Αυτή η αξιολόγηση εστιάζει σε μια πολύ σημαντική πτυχή, δηλαδή την απόφαση ε, καταλληλότητας που υιοθετήθηκε υπό το προηγούμενο πλαίσιο, δηλαδή την οδηγία του 1995 που βεβαίως προηγήθηκε του GDPR. Στη διάρκεια ε, αυτών των 20 σχεδόν ετών από την εφαρμογή της, προστα... της οδηγίας περί προστασίας δεδομένων έχουμε υιοθετήσει διάφορες αποφάσεις ε, καταλληλότητας, νομίζω 11 για διάφορες χώρες ε, όπως ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία, η Αργεντινή, για να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Και βεβαίω η συμφωνία καταλληλότητα λαμβάνεται σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και αφορά το πώς ε, εξασφαλίζεται το επίπεδο προστασίας στη συγκεκριμένη στιγμή στη συγκεκριμένη χώρα. Ορισμένες από αυτές τις συμφωνίες χρονολογούνται εδώ και αρκετά χρόνια και το GDPR απαιτεί να αξιολογήσουμε ε, κατά πόσο η ρύθμιση που είχαμε κάνει τότε ισχύει ακόμα και σωστά το ζητά αυτό. Και αυτό κάνουμε και εξετάζουμε δύο πτυχές που τις αναφέρουμε σε εσά και το Συμβούλιο. Πρώτον, τι έχει συμβεί έκτοτε, αν υπήρξαν δηλαδή νομοθετικές αλλαγές σε εκείνο το σύστημα, αν υπήρξαν συγκεκριμένες υποθέσεις, ε, εξελίξεις, πώς ε, έχει λειτουργήσει στην πράξη το σύστημα, γιατί βεβαίως δεν μας ενδιαφέρει μόνο το βιβλίο και οι κανόνες, αλλά και πώς λειτουργεί στην πράξη. Ενημέρωση λοιπόν και κατανόηση της λειτουργίας του συστήματος. Δεύτερη επιτυχή είναι να ε, ε, αξιολογήσουμε για πρώτη φορά μια επιτυχή που δεν εκτιμούσαμε όταν εγκρίθηκε η απόφαση καταλληλότητας, η οποία ανέκυψε από το δικαστήριο και συγκεκριμένα την απόφαση ΣΡΕΜΣ, δηλαδή όταν υιοθετείται μια απόφαση καταλληλότητας θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να παρακολουθήσουμε τα δεδομένα και τον κύκλο ζωής τους και όχι μόνο να αξιολογήσουμε ποια είναι η προστασία που ίσχυσε που ισχύει όταν ε, ε, τα επεξεργάζεται τα στοιχεία σε μια τρίτη χώρα μια ιδιωτική εταιρεία, αλλά και ποιες είναι οι συνθήκες ε, που ισχύουν αν οι δημόσιες αρχές της εν λόγω τρίτης χώρας έχουν πρόσβαση για λόγους επιβολής του νόμου ή εθνικής ασφάλειας. Γι' αυτό είναι φυσικά κάτι τώρα που πρέπει να συμπληρωθεί η αξιολόγησή μας με αυτές τις πτυχές. Όπως καταλαβαίνετε είναι περίπλοκο εγχείρημα, 11 χώρες και της, πολύ σημαντικές. Έχουμε κατά μέρο την Συμφωνία Καταλληλότητα Ευρωπαϊκή Ένωση Ιαπωνίας, η οποία υπόκειται σε δικό της ε, χρονοδιάγραμμα. Και αυτά είναι τα θέματα επί των οποίων πρέπει εμείς να σας κάνουμε αναφορές. Τώρα, δηλαδή κατά πόσο εξακολουθούν οι χώρες αυτές να έχουν το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας, δηλαδή αντίστοιχο με το δικό μας και αν δεν ισχύει αυτό, να προτείνουμε μέτρα ώστε να διορθωθεί η κατάσταση. Επιπλέον ασφαλιστικές δικλείδες ή και μπορεί και να πάρουμε πίσω τη συμφωνία καταλληλότητας. Αυτό θα είναι απόφαση και αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Αν χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο και ανασταλεί ισχύς, της απόφασης καταλληλότητας θα πρέπει να περάσουμε πάλι από μια διαδικασία απόφασης που προβλέπεται από το GDPR, δηλαδή γνωμοδότηση του Συμβουλίου ε, της ε, Ευρωπαϊκής Αρχής Προστασίας Δεδομένων, διαδικασία επιτροπολογίας καθώς και έλεγχος από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε καταλαβαίνετε Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, αλλά θέλουμε να ξανάρθουμε την άνοιξη με όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες για όλα αυτά τα θέματα. Και βέβαια όσο γίνεται πιο ακριβείς πληροφορίες για αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Τζιγκαρέλη για την παρουσίασή σας αυτή και αρχίζουμε τη συζήτηση με ερωτήματα των συναδέλφων. Ο συνάδελφο Μόριτζ έχει ζητήσει το λόγο και το δίνω αμέσω. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι εδώ σήμερα και για την ε, παρουσίαση, για τη δεσμότητα να απαντήσουν σε ερωτήσει. Μα Έχω μια ερώτηση, ότι η Κομισιόν διμερώς έχει διάλογο με τι εθνικέ αρχέ μεταξύ άλλων για να διαπιστωθεί ότι είναι πραγματικά ανεξάρτητες οι αρχές προστασίας δεδομένων και γίνεται λόγος για ανθρώπινους ε, οικονομικούς τεχνικούς πόρους επαρκής. Οι ανθρώπινοι πόροι σίγουρα είναι σημαντικοί, γιατί αν δεν έχουν ε, τα μέσα, οι αρχές αυτές, ο κίνδυνος είναι να πάμε πάλι στο σενάριο business as usual. Πολλές επιχειρήσεις δεν εφαρμόζουν τον νόμο ή τον ε, παραβλέπουν, γιατί δεν υπάρχει επιβολή της νομοθεσίας το Φεβρουάριο δείχνει μια έκθεση ότι η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών θέλουν περισσότερα κονδύλια για να φέρουν σε πέρα στο έργο τους ώστε να μην είναι ένας χάρτινος τίγρης ε, αυτός ο κανονισμός για την προσέγγιση των δεδομένων. Δηλαδή, χρειάζονται για παράδειγμα 37% παραπάνω κονδύλια για κάποιες χώρες 53 ή και 93, η Ρουμανία για παράδειγμα όλα τα κρατημέλη λέει θα φροντίσουν οι αρχέ σα δεδομένων να έχουν επαρκή μέσα και πόρου για να μπορούν να φέρουν πέρα στα καθήκοντά του και να ασκήσουν ε, τι εξουσίε. Του Η Κομισιόν θεωρεί ότι αρκεί ο διάλογο με αυτά τα κρατημέλη πότε θα κινήσει η διαδικασία παραβάσεις σε βάρος των κρατών μελών που αρνούνται απλά να δώσουν τους απαραίτητους πόρους στις αρχές προστασίας δεδομένων. Και αν αυτό δεν γίνει, δηλαδή η διαδικασία παραβάση πριν την αναθεώρηση του 2020, στην αξιολόγηση και στη σχετική έκθεση κομισιών θα περιλάβει την αξιολόγησή της ε, για την ανάγκη σε ανθρώπινους ε, σπόρους, ε, τεχνικούς κτλ. ώστε να ξέρουμε τι μας πρόκειται και τι χρειάζεται. Thank you. Thank you for... Ευχαριστούμε για την ερώτηση. Τονίσαμε το θέμα των πόγων ήδη από την αρχή. Με τρεις ανακοινώσεις που έχουμε διατυπώσει και δημοσιεύσει για τον κανονισμό προστασίας Κυρία Γιούροβα, έγραψε σε όλους τους υπουργούς και το υπογράμμισε αυτό το θέμα. Τι βλέπουμε. Σε πολλές περιπτώσεις δίνονται πόροι παραπάνω στις αρχές προστασίας δεδομένων. Όλοι θα θέλουν περισσότερους πόρους. Αυτό το περιμένουμε. Το θέμα είναι πιο πολύ οι ανισορροπίες που βλέπουμε να υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών. Ιταλία. 170 είναι το τελευταίο στοιχείο που έχουμε. Κάτι αντίστοιχο με το νούμερο για τη Γαλλία. Και αν το συγκρίνετε με τον πληθυσμό, με το ΕΠ και τα λοιπά, Νομίζω ότι σχετικά λιγότερα είναι τα άτομα. Είναι δύσκολο όμως να γίνει μια σύγκριση έτσι απλή, γιατί κάποιες αρχές προστασίας δομένων έχουν και άλλα καθήκοντα πέραν αυτών που άπτονται του κανονισμού προστασίας δομένων. Η Ιρλανδία είναι ένα παράδειγμα που έχει και πολλές ε, τεχνολογικές εταιρείες ή το Λουξεμβούργο με μεγάλες επίσης επιχειρήσεις εκεί. Άρα δεν είναι εύκολο να γίνει αυτή η εκτίμηση. Και αυτοί που παραπονούνται δεν είναι και κατά ανάγκη αυτοί που έχουν τα περισσότερα προβλήματα, για να το θέσω έτσι. Εμείς όμως, σε όλες τις διμερείς επαφές που έχουμε, το τονίζουμε. Θα το πούμε και στην ανακοίνωσή μας. Στείλαμε ερωτηματολόγια και σε αρχές προστασίας δεδομένων, για να μας πούν τι πόρους έχουν και τι πόρους χρειάζονται. Είναι σημαντικό το στοιχείο και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πρώτη προτεραιότητα για εμάς η ανεξαρτησία και η πόρη των αρχών προστασίας δεδομένων. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσει από του συναδέλφου. Έχω εγώ λοιπόν δύο ερωτήσει ε, έτσι γρήγορε. Λοιπόν, το ερώτημά μου σχετίζεται με αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφος και εσείς κύριε Νικόλ για το θέμα τη συνέχεια αυτής της αναθεώρησης η οποία βεβαίως δεν σημαίνει ότι θα ξανανοίξει η αξιολόγηση απλά θα παρακολουθείτε την εφαρμογή για να υπάρχει μια μεγαλύτερη συνοχή. Είπατε στην αρχή ότι μια χώρα ακόμα δεν έχει εγκρίνει συγκεκριμένη νομοθεσία οι άλλες χώρες έχουν κάποιες ε, διαφορές. Το είπε και ο συναδελφός σας. Ερωτώ λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούν να κάνουν οι χώρες και οι Κομισιόν και εμείς στο ευρωπαϊκό επίπεδο για να δημιουργηθεί αυτή η μεγαλύτερη συνοχή στην εφαρμογή του GDPR στις χώρες μας. Μετά μια ερώτηση και για τον κύριο Τζενκαρέλη, αλλά θα την κάνω μετά. Ναι. Απαντήστε πρώτα εσείς, παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι, είναι προφανές από την ε, ανακοίνωση που βγάλαμε τον Μάιο που έχουμε τα όσα μας λέει ο κλάδος ε, και η κοινωνία των πολιτών ότι το θέμα της συνοχής της εφαρμογής είναι πάρα πολύ βασικό και εδώ πέρα πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ των διαφορετικών καταστάσεων. Ο κανονισμός αφήνει ένα περιθώριο λιγμών στα κράτη-μέλη. Ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι η ηλικία συνένεσης ε, για τις ψηφιακές υπηρεσίες και μετά τα κράτη-μέλη θα χρησιμοποιήσουν αυτήν την ε, ευελιξία, αυτό το περιθώριο και στο μέλλον πιθανότατα όταν θα αναθεωρηθεί ο κανονισμός θα έχουμε ένα στοιχείο ευελιξίας στο οποίο θα επανέλθουμε. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Οπότε εδώ πέρα μπορούμε πραγματικά να πιέσουμε για να μειωθεί ο κατακαιρματισμός που υπάρχει στον γενικό κανονισμό. Από την άλλη, από την άλλη υπάρχει εκεί όπου υπάρχει απόκληση που δεν είναι εντός ε, του πλαισίου που υπάρχει ερχόμαστε σε συνεννόηση με τα κράτη-μέλη για να μας ξεκαθαρίσουν πώς έχουν οι νόμοι η σχετική. Και έχουμε εδώ πέρα διάφορα μηνύματα ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα εκεί όπου δεν υπάρχει περιθώριο λιγμών. Οπότε αυτό είναι θέμα νομοθεσίας. Αλλά υπάρχει μετά άλλο ένα κομμάτι το οποίο αφορά την εφαρμογή και τις συμβουλές των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων. Και βεβαίω, αν πάνε σε διαφορετικέ αρχέ προστασία δεδομένων, του λένε άλλα πράγματα καμιά φορά. Αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα και νομική αβεβαιότητα. Ε, Ακριβώ εδώ πέρα λοιπόν χρειάζεται κατεύθυνση όχι σε εθνικό αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. για να δούμε πώς αντιμετωπίζονται συγκεκριμένα ζητήματα. Υπάρχουν ήδη 24 κατευθυντήριες γραμμές, πρέπει να ζητήσουμε περισσότερες και να ενθαρρύνουμε αυτό το οποίο είπα πριν, τον κώδικα συμπεριφοράς. Γιατί άπαξ υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για έναν κλάδο, π.χ. τις μεταφορές, τότε θα επικυρωθεί τροποντινά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχών Σοπικών Δεδομένων. Και θα λένε ότι σε αυτόν τον κλάδο έτσι εφαρμόζουμε, έτσι αντιλαμβανόμαστε αυτήν την ε, πολιτική. Και αυτό βεβαίως θα μας βοηθήσει, θα βοηθήσει ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε αυτά θα γίνουν για να υπάρξει μια πιο ομοιόμορφη εφαρμογή. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ. Τώρα θα δώσουμε τον λόγο στον κύριο Τσενκαρέλη που θα μας μιλήσει για τη διεθνή διάσταση. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο με απασχολεί ιδιαιτέρως ως Ιταλίδα. Η συνεργασία δηλαδή μεταξύ των αρχών που είναι πάντα πολύ σημαντική. Μιλήσατε λοιπόν για συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει ακόμα για να βελτιωθεί αυτή η συνεργασία. Που ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Εσείς αναφέρατε παραδείγματος χάρη τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου που αναπτύσσεται και εξελίσσεται και βεβαίως ε, η προστασία των δεδομένων έχει τεράστια σημασία. Οπότε, σας ερωτώ, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε, πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τη συνεργασία μεταξύ των αρχών που ασχολούνται με την προστασία των δεδομένων στο διεθνές επίπεδο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή η οποία για ε μας είναι από τις ε, σημαντικότερες ε, και αφορά επίσης το πώς η προστασία των δεδομένων θα πάει από τα βιβλία στην πράξη. Είναι η άλλη όψη του νομίσματος, δηλαδή να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή πρώτα στην Ευρώπη αλλά και παρά έξω. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία. Μας διευκολύνει λοιπόν το να έχουμε κοινού ε, κανόνες ε, και στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης, ε, στον τομέα της εφαρμογής του ποινικού δικαίου, το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά Δηλαδή, αν δύο εισαγγελεί πρέπει να συνεννοηθούν σε διαφορετικέ χώρε, αν έχουν κοινού κανόνε, μπορεί να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών και να προχωρήσουν κοινέ έρευνε. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Λοιπόν, εμεί θεωρούμε ότι αυτή η σύγκληση που αναφέραμε στο επίπεδο των κανόνων ε, το βοηθάει αυτό. Θεωρούμε επίσης ότι υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση γιατί απέναντι σε γίγαντες έχουμε τις αρχές ε, προστασίας δεδομένων της δικές μας και άλλων χωρών οι οποίες ε, αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Επίσης ε, βλέπουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για εμάς, ότι σε χώρες π.χ. της Λατινικής Αμερικής οργανώνται σε περιφερειακό επίπεδο. Εμείς βεβαίως ε, ε, είμαστε συνηθισμένοι να δουλεύουμε έτσι. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Αλλά ακριβώς θέλουμε να διευκολύνουμε την συνεργασία γιατί θα μπορούσαμε έτσι να έχουμε έναν πολλαπλασιαστή. Και το δίκτυο αυτό το λατινοαμερικάνικο ή ιβυροαμερικάνικο θα μπορούσε να έχει κάποια συγκεκριμένη λειτουργία. Τι κάνουμε λοιπόν. Ο Γενικός Κανονισμός μας δίνει την δυνατότητα στην Κομισιόν εννοώ να διαπραγματεύεται διεθνείς ε, συμφωνίες εστιάζοντας στην ε, συνεργασία ε, αυτή και έχουμε πει στο Συμβούλιο Προστασία Δεδομένων, να μα πει ποιε θα είναι οι χώρε προτεραιότητα. Αυτό όμω είναι μέσω μακροπρόθεσμο. Αυτό το οποίο κάνουμε άμεσα είναι να δημιουργήσουμε αυτό το οποίο λέμε μια ακαδημία προστασίας δεδομένων που θα φέρει τις αρχές προστασίας δεδομένων της Ευρώπης ε, ε, και θα προσκαλέσει τις αρχές μας να ανταλλάξουν βέλτιστες ε, πρακτικές και εμπειρίες και να αναπτύξουν κοινά εργαλεία ερμηνείας της νομοθεσίας. Αυτό έτσι ως αφετηρία από κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε βασικό, αλλά όπως γνωρίζουμε, η εμπειρία του ότι ξέρουμε ποιο, σε ποιον να τηλεφωνήσουμε και με ποιον να ανταλλάξουμε πληροφορίες είναι πάρα πολύ σημαντική. Τότε έχουμε αυτή τη μία πτυχή, δηλαδή του πώς λειτουργούν οι αρχές προστασίας δεδομένων. Η άλλη πτυχή, γιατί βεβαίω πρέπει να είναι διμερές ε, το θέμα αυτό, είναι οι δικές μας οι αρχές ε, να έχουν ε, ένα μέρος όπου θα μπορούν να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να συνεργάζονται. Κάτι πολύ συγκεκριμένο λοιπόν. τώρα τα έχουμε στήσει, και θα είναι έτοιμα τους επόμενους ε, μήνες. Ελπίζω να απάντησα. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί κύριοι για την παρουσίαση αυτή. για την διαδικασία αξιολόγησης ε, του Γενικού Κανονισμού και για τις ε, πλήρεις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε και για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Διακόπτεται λοιπόν πάλι η συνεδρίαση. Το επόμενο θέμα το κάνει ο κύριος Λόπες Αγγιλιάρα. Ευχαριστώ, Thank you. for remaining faithful. Σας ευχαριστώ που μείνατε πιστοί και παρακολουθείτε την ατζέντα τη σημερινή που τυχαίνει να, μάλιστα τώρα να είναι το τελευταίο σημείο. Τελευταία ώρα. 4.30 με 5.30. Θα ακολουθήσουμε τις πληροφορίες από το Συμβούλιο προς το Κοινοβούλιο για την πρόσφατη ε, πρόταση για το άρθρο 7 για την κατάσταση δικαίου, ε, του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία. Φαντάζομαι όλοι γνωρίζετε τα σχετικά και σήμερα θα ακούσουμε άμεσα από το Συμβούλιο το οποίο εκπροσωπεί εδώ η Φιλανδική ε, Προεδρία, ο Φιλανδός πρέσβης στην Ένωση που θα μας πει τι συμβαίνει με το άρθρο αυτό για την Ουγγαρία. Είμαι βέβαιος πως το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει ε, μπορεί να μην μπορεί να υπάρχει νομική αντίρρηση, ένσταση, α, α, μπορεί να μην υπάρχει νομική υποχρέωση ε, λόγω του και ένσταση ε, να ακουστεί η φωνή του Κοινοβουλίου σε μια συζήτηση που συνεχίζεται όπου το Κοινοβούλιο ανέλαβε την πρωτοβουλία πρώτη φορά. Όποτε λοιπόν θα ακούσουμε την έκθεση πρόοδου, αλλά να ξε... ακούσουμε πρώτα την εκπρόσωπο του Συμβουλίου εδώ, ε, θα πρότεινα maximum 10 λεπτά για τα μέλη, ε, για να μπορέσουμε μετά να ακούσουμε και τα μέλη. Παρακαλώ, κύριε Χτιστάκη. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη βουλευτές Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρώτο Επιτροπής, τον κύριο Λόπεθ καθώς και ε, την κυρία Τέρμπο Σκορφίλτ που είναι η συγκέντρα του Ευρωκοινοβουλίου για την πρόταση περί Ουγγαρίας για την προσκλησή να έρθω εδώ και να ενημερώσω την Επιτροπή σας για το πώς έχει η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του άρθρου 7 και την Ουγγαρία. Όπως γνωρίζετε, ο τομέα αυτό το κράτο δικαίου, είναι μία από τι προτεραιότητε τη Φινλανδική Προεδρία. και πράγματι νομίζω ότι είναι προτεραιότητα συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο σεβασμό στι θεμελιώδεις αξίε είναι κάτι απολύτω αναγκαίο για να είναι αποτελεσματική, αποδεκτή και αξιόπιστη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδικασία του άρθρου 7 είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας στην εργαλειοθήκη για το κράτος δικαίου. Στη διάρκεια της Προεδρίας μας προσπαθήσαμε να προχωρήσει η συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει το... συνολικά αυτή η εργαλειοθήκη να προχωρήσει. Μεταξύ των άλλων και ο διάλογος για το κράτος δικαίου για ανταλλαγή βέλτιση των πρακτικών προληπτικών μέτρων είναι ένα εργαλείο. Νομίζω συμφωνούν όλοι πως τα θετικά προληπτικά εργαλεία θα πρέπει να προτιμώνται στο βαθμό του δυνατού. Ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι, έχουμε προχωρήσει με τις διαδικασίες του άρθρου 7. Από το πρίσμα των απόψεων των ε, περισσότερων κρατών μελών του Συμβουλίου, όπως θεωρήσαμε σκόπιμο να πράξουμε. Για την περίπτωση της Ουγγαρίας αυτό τι σήμαινε. Οργανώσαμε μια πρώτη ακρόαση στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων του Σεπτεμβρίου. Είχε περάσει σχεδόν ένας χρόνος ε, από τότε που πήραμε την πρόσφατη πρόταση του Κοινοβουλίου. Θεώρησαμε λοιπόν ότι καλό είναι να γίνει μια πρώτη ακρόαση. Η πρώτη ακρόαση αυτή ήταν γενική, δηλαδή συμπεριλάμβανε όλα τα ζητήματα και αυτά τα οποία περιλαμβάνονταν στην πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου. Επίσης δόθηκε στην Ουγγαρία δυνατότητα να ακουστεί και αυτό επίσης θα σημαντικό. Όπως ορίζουν όριο, όπω εγκρίθηκαν τον Ιούλιο από το Συμβούλιο, στι αρχέ πρώτη ακρόαση, η Φιλοδική Προεδρία ενημέρωσε εν συντομία το Συμβούλιο για τι επαφέ που είχε με το Κοινοβούλιο και τι απόψει του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο τη ετολογισμένη του πρόταση. Για την προετοιμασία αυτή τη ακρόαση ενημέρωση, οργανώθηκε άτυπη συνάντηση με τον πρόεδρο τη Λύπε και τον εισηγητή, καθώ και με τι μελλοντικέ προεδρίε, την Κροατία και τη Γερμανία. Μετά από αυτήν ε, την ε, ενημέρωση στο Συμβούλιο, η Ουγγαρία κλήθη να παρουσιάσει τις απόψεις της ε, για την έκθεση του Κοινοβουλίου συνολικά. Διότι πρέπει να ακούγεται το κράτος μέλος που το αφορά η διαδικασία του άρθρου 7. Αυτό είναι σαφές και το λέει η διαδικασία του άρθρου 7 στην παράγραφο 1. Επίση αυτοί οι όροι που εγκρίναμε το καλοκαίρι ορίζουν ότι θα πρέπει να δοθεί επαρκή χρόνος για τον λογοκράτο, ώστε να εξηγήσει τη θέση του στην πρώτη ακρόαση. Μετά την ακρόαση τα άλλα κρατημέλη είχαν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις, μάλλον στο τέλος της ακρόασης. Ετέθησαν τα εξή. Ακαδημαϊκή ελευθερία, ελευθεροτυπία, διαφθορά, ελευθερία έκφρασης, ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, της δικαιοσύνης. Χαίρομαι πολύ που μπορώ να σας πω ότι έγινε επικοδομητικά, μια επικοδομητική ακρόαση και στο τέλος της συζήτησης ε, η Προεδρία κατέληξε σε, μια, σε ένα διαδικαστικό συμπέρασμα, ότι δηλαδή θα πρέπει να συνεχίσει να επιλαμβάνεται το θέμα στο Συμβούλιο. Ποιε είναι τώρα οι επόμενες εξελίξεις. Η Κορεπέρα αποφάσισε χθες να γίνει μια δεύτερη ακρόαση με την Ουγγαρία στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 10ης Δεκεμβρίου. Η ακρόαση αυτή θα προετοιμαστεί έτσι πιο αδιεξοδικά στην κορυφή της επόμενης εβδομάδας. Και αυτή τη φορά θα προτείνει η Προεδρία μια θεματική ακρόαση. Κορεπέρ θα διαλέξει λίγα βασικά ζητήματα για αυτήν την ακρόαση, ώστε να γίνει μια πιο ουσιαστική σε βάθος συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα τέλος να πω πως η Φιλανδική Προεδρία συμφωνεί πως το Συμβούλιο θα πρέπει να τηρείται ενήμερο για τις απόψεις του Κοινοβουλίου σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, διότι πρόκειται και για μια διαδικασία που το ίδιο το Κοινοβούλιο δρομολόγησε. Χαίρομαι που θα μπορέσω να ακούσω σήμερα τις απόψεις ε, της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, τις οποίες και θα μεταφέρω βέβαια στην επόμενη ακρόαση που θα οργανώσει το Συμβούλιο. Επομένως, κυρίε και κύριοι, αυτά είναι τα, ε, έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι τώρα. Έχουν γίνει υποδομικές συζητήσεις και έτσι ελπίζουμε με αυτό το πνεύμα δηλαδή να συνεχίσουμε, πάντοτε βέβαια με την πεποίθηση πως το κράτος δικαίου τελικά είναι κάτι το οποίο ενώνει τα κράτη-μέλη της Ένωσης και τους πολίτες της. Θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά την Επιτροπή σας και ιδίως ε, τον κύριο Λόπεθ Γιλάρ και την κυρία Τελμποσκόρφιλτ για την καλή συνεργασία που είχαμε. Και βεβαίως είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ζησλάκη. Να ακούσουμε πρώτα, θα έλεγα, τον αρμόδιο εισηγητή. Την εισηγητή, την Ντελμπο Κορφίλτ. Ντελμπό Κορφίλτ, έτσι δεν σας λένε. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Για πόσο να πω, τρία-πέντε λεπτά. Για να, έχει χρόνο, να έχουν χρόνο και άλλοι Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή Λίμπε σας ευχαριστώ που είστε εδώ, ε, την Φιλανδική Προεδρία και σας ευχαριστώ όχι μόνο γιατί είστε μόνο σήμερα εδώ, σας ευχαριστώ γιατί, κυρίως για τη δουλειά που έχετε κάνει εδώ και πολλούς μήνες και δεν είναι κάτι το τυπικό από πλευρά μου. Νομίζω πως όλοι μπορούμε, όλοι οι προβλεφτές μπορούμε να σας ευχαριστήσουμε. Η κοινωνία των πολιτών στην Ουγγαρία, τα κοινοβούλια των άλλων χωρών αλλά και τα κρατημέλη γιατί αποδείξατε ότι δείξατε μεγάλη σοφία, θάρρος, και τα μετράω τα λόγια μου γιατί δεν ήταν προφανές να αναλάβετε αυτή την υπόθεση όταν αναλάβατε την Προεδρία γιατί είχε θαυτεί κατά κάποιο τρόπο το Συμβούλιο. Δεν είχε απαντήσει καν στο Κοινοβούλιο το Ευρωκοινοβούλιο είχε το θάρρο να υπερψηφίσει αυτή την έκθεση και είχε μείνει χωρίς απάντηση. Οι επίτροποι έκαναν τη δουλειά του. Εσεί μπορέσατε να δράσετε, να ενεργήσετε γρήγορα και αποτελεσματικά, αλλά και με μεγάλη ε, ευφυα, εξισορροπώντα του διάφορου ε, παράγοντε αυτού του ε, θέματο, γιατί δεν είναι άνετη η κατάσταση, δεν είναι ομοσπονδιακή η Ευρώπη, είναι διακυβερνητική. Οι αποφάσει λαμβάνονται ομόφωνα και για τα κράτη-μέλη να κρίνουν έναν δικό τους είναι πολύ δύσκολο. Αυτή η ακρόαση λοιπόν είναι πραγματικά ε, ε, πρεμιέρα. Όταν ε, Βέβαια, ενεργοποιήθηκε το άρθρο 7, ήταν πάλι πρεμιέρα και χρειάστηκε μεγάλη διπλωματία, πολιτική λεπτότητα και θάρρος. Ε, πετύχατε δεύτερη ακρόαση το Δεκέμβριο. Ξέρω ότι σε διάφορες φάσεις η συνεργασία μας τους τελευταίους μήνες ανησυχήσατε ότι δεν θα μπορούσατε να τα καταφέρατε και νομίζω πως ήταν εξαιρετικό το νέο ε, και πάλι μπράβο σας. Μένει ένα δύσκολο σημείο ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει βρει ακόμα τη θέση του σε αυτή τη διαδικασία. Η διάσταση ή δια... θεσμική είναι ελαττωματική από αυτή την άποψη. Ε, να θυμίσω το άρθρο 13 παράγραφος 2. Είναι σημαντικό να το λέμε ότι κάθε θεσμός ε, ενεργεί μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του όπως προβλέπονται από τη συνθήκη σύμφωνα με τις διαδικασίες, του όρους και τον τρόπο με τον οποίο ε, προβλέπεται στις συνθήκες και ενεργούν μεταξύ τους με πιστό τρόπο και θεμητό τρόπο. Εδώ όμως δεν υπάρχει θεμητή συνεργασία γιατί το άρθρο 7 το οποίο ενεργοποιήθηκε για την Πολωνία είναι παρούσα παντού σε όλες τις ακροάσεις και όλα τα στάδια της διαδικασίας, ενώ εδώ όχι. Πιστεύω πως είναι κρίμα. Είναι κρίμα από θεσμική άποψη, είναι κρίμα α, όσον αφορά το σεβασμό του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί κάποιες φορές αισθανόμαστε προσβεβλημένοι ως Ευρωβουλευτές, αλλά είναι και κρίμα γιατί εδώ μέσω εμού, αλλά και μέσω του κυρίου Λόμπες Αγγιλάρ, Προέδρου της Επιτροπής Λίμπε και άλλων ερετών, εδώ έχουμε κάνει τρομερή δουλειά εδώ και ε, μία δεκαετία στο Κοινοβούλιο έχουμε εμπειρογνωμοσύνη και ε, Εάν μπορούσαμε ευρύτερα να το χρησιμοποιήσουμε στη διάρκεια των συμβουλίων και μέσα στις ακροάσεις, θα μπορούσαμε σίγουρα να κάνουμε ε, πρόοδο και να κατανοήσουμε καλύτερα τα πράγματα και να τα καταστήσουμε κατανοητά για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Οπότε είναι μια δουλειά που πρέπει να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ελπίζω, ξέρω πως το προσπαθήσατε, ελπίζω πως και άλλοι θα το προσπαθήσουν μετά από εσά. Ξέρω επίση ότι το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει απέρα ακόμα περισσότερο να αγωνιστεί, αλλά να συμμετέχει και με καλύτερο τρόπο σε αυτή τη διαδικασία, η οποία θα συνεχιστεί με τη δεύτερη ακρόαση το Δεκέμβριο. Δεν θα σταματήσει όμω εκεί, γιατί βέβαια η κατάσταση δεν έχει ρυθμιστεί στην Ουγγαρία για διάφορα ζητήματα. Ελπίζω πω η Προεδρία, η Κροατική και η Γερμανική με τη σειρά του θα ασχοληθούν με αυτό το θέμα με την ίδια σοβαρότητα που το κάνατε και εσείς. Ελπίζω επίσης ότι η εργασία επί της οποίας δεσμεύτηκαν οι Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για να προχωρήσουμε για την εγκαθίδρυση μηχανισμών κράτους δικαίου, μιλήσατε για πρόληψη. Ναι, είχετε δίκιο ότι έπρεπε να έχει υπάρξει πρόληψη νωρίτερα, όμως τώρα υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες. Έχουμε ένα πρόβλημα με το άρθρο 7 και όπως εμείς το ενεργοποιήσαμε δεν υπάρχει πλαίσιο, δεν υπάρχει χρονικό πλαίσιο, δεν ξέρουμε πότε θα σταματήσει η διαδικασία, δεν προβλέπονται κυρώσεις και δεν υπάρχει ούτε μέθοδος. Εμείς ε, εφευρίσκουμε από την πλευρά σα εσείς και εμείς από τη δικιά μας. Αλλά θα πρέπει να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις διαδικασίε ώστε πάντοτε να έχουμε τις βάσεις, τις απαραίτητες που είναι ε, ε, για τη δημοκρατία γιατί αν δεν υπάρχει η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, αν δεν ισχύει η δημοκρατία στα κράτη-μέλη τη ε, ε, πλήρω. Οι Ευρωβουλευτέ που είναι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών και τη κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να συμμετέχουν ακόμη περισσότερο. Εδώ και 14 μήνες ψηφίστηκε η έκθεση αυτή. Από τα δύο τρίτα τη Ολομέλεια, το είπα ήδη. Ήταν ήδη μεγάλη απόδειξη παρησία από πλευρά αυτού του Κοινοβουλίου γιατί ε, Πολλοί μάλιστα ήταν μέλη του ίδια ομάδα ε, στην οποία ανήκει και το κόμμα τη Ουγγρική κυβέρνηση. Το Συμβούλιο έκανε την πρώτη του ακρόαση σχεδόν ένα χρόνο μετά από την υιοθέτηση. Στις 16 Σεπτεμβρίου και στις 10 Δεκεμβρίου θα γίνει η επόμενη ακρόαση. Και εδώ και χρόνια η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται για πολλά πολλά ε, θέματα. Πολύ πρόσφατα τη Δευτέρα, την περασμένη, το άνοιγμα της, του Πανεπιστημίου της Κεντρικής Ευρώπης ε, ε, στην Ευρώπη, στην ε, Βιέννη με συγχωρείτε, δείχνει πως η κατάσταση συνεχίζεται. Αυτή η κατάσταση στην Ουγγαρία που για πολλά σημεία δεν έχει βελτιωθεί, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ανεξαρτησία των ακαδημαϊκών ε, ιδρυμάτων, η κατάσταση για τους μετανάστες μας οδηγούν, μας, μας είναι σημαντικά για όλους μας, όχι μόνο για την ε, Ουγγαρία, γιατί το ντόμινο, το εφεντόμινο μπορεί να λειτουργήσει και γιατί η Ουγγαρία στο Συμβούλιο μπλοκάρει την πρόοδο για άλλα θέματα. Και εδώ κυρίως είναι πραγματικά κρίμα που το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να προχωρήσει για τις προτάσεις που έγιναν για μια ετήσια έκθεση για το κράτος δικαιού στις χώρες δεν έχει μπορέσει να προχωρήσει και για διάφορες προτάσεις του το Συμβουλίου για να προχωρήσει το θέμα του μηχανισμού για το κράτος δικαίου. Η Πολωνία και η Ουγγαρία μπλοκάρουν κάθε φορά και πρέπει να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό για να έχουμε υγιές μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Τώρα προτείνω να ακούσουμε τους σκιώδεις που είναι παρόντες στην αίθουσα. Κυρία Πουρέκ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι οι εξελίξεις στην Ουγγαρία είναι ενισχυτικές Η συνάδελφος από τους πράσινους τα είπε ήδη. Μετά από 25 χρόνια λειτουργία στην Βουδαπέστη του Κέντρο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο αναγκάστηκε να φύγει από την χώρα και να πάει στην Αυστρία. Και η Ουγγρική κυβέρνηση δεν κύρωσε την συμφωνία που θα επέτρεπε να συνεχίζει ε, την λειτουργία του με βάση το νόμο του 2017 για τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέτασε το θέμα αυτό από τις εκλογές του 2010, πέρασε το Κοινοβούλιο πέντε ψηφίσματα, κάτι το οποίο δεν απέδωσε. Γι' αυτό η κυρία Σαρτζεντίνη ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2017 να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 Έκτοτε όμως ε, το Συμβούλιο δεν ακολούθησε τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, αλλά τώρα, και εδώ πέρα έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του ότι το άρθρο 7 δεν είναι αποτελεσματικό, ε, πρέπει να δούμε ότι υπάρχει σαφής ανάγκη ενός παράλληλου μηχανισμού. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι στηρίζω πλήρως την πρωτοβουλία να ζητηθεί γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια. Όπως είχα προτείνει και εγώ ως και Σας ευχαριστώ. Από το Ρινιού η σκιώδηση συγκεκριά επίσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Φιλανδική Προεδρία για τις ενεργειές της. Ελπίζω ότι αυτή η δυναμική θα συνεχιστεί με τη δεύτερη ακρόαση που έχει προγραμματιστεί για το Δεκέμβριο και παραπέρα επί Κροατικής Προεδρίας. Ως και ηγετρία της ομάδας Ενιού, πρέπει να εκφράσω την απογοήτευσή μου για το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο για πρώτη φορά κίνησε την διαδικασία άρθρο 7 για την Ουγγαρία, δεν είχε το δικαίωμα να λάβει μέρος στην ακρόαση αυτή ενώπιον του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Άκουσα τα επιχείρηματα του Συμβουλίου ότι δεν προβλέπεται η συμμετοχή του Κοινοβουλίου ούτε από την συνθήκη ούτε από τον κανονισμό του Συμβουλίου. Δεν ε, με πείθει εμένα αυτό. Εξάλλου υπάρχει προηγούμενο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ας πούμε, συμμετέχει σε κάποιε συνεδρίες του Συμβουλίου. Ελπίζω λοιπόν να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τη γνωμοδότηση που ζητήσαμε από την νομική μας υπηρεσία και θέλω να επανέλθω σε αυτό το οποίο είπε η συνάδελφος. Για το άρθρο 13 που ζητάει από όλα τα θεσμικά όργανα να συνεργάζονται. Η θέση του Κοινοβουλίου είναι γνωστή και είχε τεκμηριωθεί στο ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2018. Νομίζω ότι είναι ε, σοβαρός λόγος ανησυχίας γιατί εδώ πέρα επαβαθμίζεται η αξιοπιστία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αν οι παραβιάσεις των αξιών της Ένωσης είναι κατόπιο παίρνουμε Επίσης, αυτό δεν σταμάτησε την επιστοχώρηση του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία και, για να είμαι ειλικρινής, ενώ εμείς έχουμε κολλήσει στα διαδικαστικά, Σχεδόν κάθε μέρα ακούμε διάφορα πράγματα για την πίεση που ασκείται στους δημοσιογράφους, μείωση της ελευθερίας των ΜΜΕ. Ή για το ότι δεν υπάρχει χώρος για την κοινωνία των πολιτών. Όπως ακούσαμε σήμερα και από την ε, εκδήλωση που οργάνωσε η συγκεκριά. Ενώ λοιπόν έχουμε κολλήσει στα διαδικαστικά ε, γίνεται επιδρομή στα γραφεία των συναδέλφων μου από το Momentum και αν θυμάμαι καλά οι συνάδελφοί μου ήταν εκεί και κάποιος είπε ότι ο μόνος χώρος που υπάρχει για τα ΜΜΕ και την κοινωνία των πολιτών για να εκφραστούν ελεύθερα στην Ουγγαρία είναι τα δικαστήρια. Μόνο εκεί μπορεί να μιλήσουν ελεύθερα για το τι συμβαίνει. και βεβαίως ε, εγείρονται και οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία να διατηρήσουμε την πίεση στην ευρική κυβέρνηση και να σταματήσει συστηματική επίθεση στις αξίες της Ένωσης. Η ερώτησή μου λοιπόν επιτέλους είναι η εξή. Πώς βλέπετε να προχωράει αυτό το θέμα. Και δεύτερον, είδα την απάντηση της Φιλανδικής Προεδρίας στον κύριο Σασόλη αντιλαμβάνομαι ότι για την ώρα δεν υπάρχει ε, θέση για εμάς στην ακρόαση του Δεκεμβρίου. Ε, μπορούν να περιληφθούν οι προτάσεις μας στην ημερήσια διάταξη της ακρόασης. Γιατί μπορούμε να κάνουμε τέτοιες προτάσεις. Και υπάρχει χώρος για να παρουσιαστεί ένα έγγραφο για τις ιδέες μας για το τι πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ζλάκη, να ολοκληρώσουμε με τον κατάλογο των βουλευτών και μετά να μας τα πείτε εσείς, αν συμφωνείτε. Θέλετε. Έτσι. Κύριε Χιτβέγγε. Ευχαριστώ, θα μιλήσω γκρικά κύριε Πρόεδρε. Η Ουγγαρία δεν έχει πρόβλημα με το κράτος δικαίου. Σε καμία περίπτωση. Το κράτο δικαίου είναι το θεμέλιο τη δημοκρατία μα και τη συμμετοχή μα στην Ένωση. Έχουμε ένα πρόβλημα με το γεγονό ότι αυτό το χρησιμοποιούν για όπλο εναντίον μα, ω όπλο εναντίον μα υπάρχει παρερμηνία ε, και πολιτική μεροληψία. Είναι μια πολιτική επίθεση από τη φιλελεύθερη αριστερά. Οι πιο πολλοί Ούγγροι θεωρούν ότι η χώρα δέχεται συνεχώς επίθεση. Μόνο και μόνο επειδή δεν θέλουν να πάρουν μετανάστες. Και επειδή θέλουμε να, να υποστηρίξουμε τη χριστιανική μας παράδοση, μεταξύ άλλων. Δηλαδή μας κατηγορούν και θεωρούν ότι εμείς φταίμε για πολλά πράγματα το Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διεξάγει με τέτοια διαδικασία. Αυτό προβλέπεται από την νομοθεσία. Όμω οι αριστεροί, οι φιλελεύθεροι βουλευτέ θέλουν η Επιτροπή αυτή εδώ να συμμετέχει ενεργά. Αυτό παραβιάζει το εφιστάμενο δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο. Δεν έχει πλέον κανένα ρόλο και είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Κύριε Ινσυρή, λέω να πάρει δεύτερη το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τη Φιλανδική Προεδρία καθώς και τους εισηγητέ μας. Το ερώτημά μου ουσιαστικά είναι ποιο είναι το επόμενο ε, βήμα. Ε, είπατε ότι έχετε και δεύτερη ακρόαση. Συγκεκριμένα τι συζητήθηκε, ποιοι είναι οι τρόποι να προχωρήσουν αυτές οι συζητήσεις. Ξέρουμε πολύ καλά, παρά τα όσα ε, είπε ο συνάδελφος από το Φιντές, ότι ο Ούγγρος Πρωθυπουργό Όρμπαν ε, ε, ουσιαστικά καταστρέφει τη δημοκρατία, παραβιάζει το κράτος δικαίου και θα έλεγα και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής παραβιάζει. Τα θεμελιώδη δικαιώματα για να είμαι πιο συγκεκριμένη. Με βάση το Freedom House και το δημοκρατικό του δίκτυ, σήμερα έχουμε στην Ένωση μια ανελεύθερη δημοκρατία. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε μηχανισμούς, ισχυρούς μηχανισμούς, ώστε όλα τα κράτη-μέλη να συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα όταν προσχωρούν στην Ένωση. Όμως, δυστυχώς, δεν έχουμε ένα τόσο ισχυρό μηχανισμό ε, που να ισχύει για όταν γίνουν. Δηλαδή, αφού προσχωρήσουν, δεν είναι τόσο ισχυρό ο όσο είναι πριν προσχωρήσουν. Εμείς θέλουμε την αρχή της αιρεσιμότητας να συνδεθεί με τον προϋπολογισμό. Πώς προχωρούν οι συζητήσεις στο Συμβούλιο σε ό,τι αφορά το σημείο αυτό. Είναι έτοιμο, αν χρειαστεί το Συμβούλιο, πώς προχωρούν οι συζητήσεις τουλάχιστον μέχρι τώρα, να χρησιμοποιήσει το μηχανισμό της ειδικής πλειοψηφίας για να πέσει για μια αρχή ερεσιμότητας, αν δεν συμφωνεί, κυβέρνηση Φιντέ τη Ουγγαρία. Είναι απαράδεκτο να παίρνει δισεκατομμύρια ευρώ ενώ ταυτόχρονα η Ουγγαρία παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα διαλύει τη δημοκρατία και δεν τηρεί τις βασικές θεμελιώδεις μας αρχές και αξίες. Ευχαριστώ. Κυρία Ντόμπρεφ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γκρικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα θέλω να θέσω ένα ερώτημα που θα θέσαν πολλοί συνάδελφοι, αν έχει αλλάξει κατάσταση στην Ουγγαρία πρόσφατα. Στις 13 Οκτωβρίου έγιναν τοπικές εκλογές και ο κύριος Όρμπαν ιτήθηκε. Τέθηκε το ερώτημα, μπορεί να αλλάξει. Θα αναγνωρίσει ότι αυτή η πολιτική μίσους καταστρέφει την Ουγγαρία. Αυτό μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι για λίγες μέρες το πιστέψαμε. Επειδή είπε ωραία λόγια για τη δημοκρατία, ότι θα δεχθεί τη βούληση του λαού, κάλεσε και τον δήμαρχο της αντιπολίτευσης το Δήμαρχο της Βουδαπέστης ε, σε μια συνάντηση. Ο μόλις έφυγε από το γραφείο του, τον μαχαίρωσε πισόπλατα και προσπαθεί να ξαναπάρει ε, τις εξουσίες από τους Δήμους. Ε, προσπαθεί να κόψει τους ε, πόρους που, που να περιορίσει τις ελευθερίες τους. Ταυτόχρονα περιορίζει και τον ρόλο των δημοσιογράφων. Οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν καν να μπουν στο κοινοβούλιο για να κάνουν τη δουλειά του. Είναι ένα πολύ αρνητικό προηγούμενο στην ιστορία της δημοκρατίας. Και αν θέλετε να καταλάβετε τον Ορμπάν και την κυβέρνησή του, σας πω το εξή. Από τη στιγμή που ενεκρίθη ο πρώτος ε, ο νέος Ούγκρος Επίτροπος, την επόμενη μέρα κατέθεσε η κυβέρνηση νομοσχέδιο για αλλαγή των δικαστηρίων. Δεν είχε υποσχεθεί ότι όχι ποτέ τα διοικητικά δικαστήρια σε αυτό το σύστημα δεν θα αλλάξουν κτλ. κτλ. Γιατί πρέπει να τηρήσουμε τα ενωσιακά πρότυπα. Ορίστε που τώρα κατέθεσαν αυτό το νομοσχέδιο, αλλά με διαφορετικά, διαφορετικές διατάξεις που θα επιτύχει όμως ακριβώς τον ίδιο σκόπο. Όλα τα δικαστήρια, ακόμη και το ανώτατο δικαστήριο, θα είναι πλέον υπό την επιρροή του κυρίου Όρμπαν και αυτό λίγες εβδομάδες μετά τις τοπικές εκλογές. Πραγματικά εξεπλάγει βλέποντα να λέει το κυβερνών κόμμα, όχι, όχι, όχι, το κράτο δικαίου είναι ε, μια χαρά στην Ουγγαρία, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να αναλύει την κατάσταση και τους ε, ε πρόκειψε μια νέα ιδέα. Μα δεν υπάρχει ε, ιδέα ε, του κράτους δικαίου. Τι να αναλύσει κανεί. Δεν υπάρχει κάτι να αναλύσει κανεί. Η Ουγγαρία δεν ανήκει στην ε, κοινότητα των δημοκρατικών κρατών που σέβονται το κράτος δικαίου. Αυτό που θέλω να σας πω είναι παρακαλώ μην αφήσετε τον κύριο Όρμπαν να σας εξαπατήσει και να σας εξαπατά συνεχώς. Εδώ και μια δεκαετία παίζει αυτά τα παιχνίδια. Εμείς στην Ουγγαρία αγωνιζόμαστε για να πάψει ο Όρπα να εξαπατά τους Ούγγρους πολίτες. Δεν πρέπει να τον πιστέψετε. Δεν είναι πρόβατο, είναι λύκος που φοράει μία ε, προβιά και καταλύει τη δημοκρατία. Ευχαριστώ. Euh, euh, Έχω μια ερώτηση σε σχέση με την κατάσταση των ΜΚΟ στην Ουγγαρία. Τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να στραφεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με προσφυγή κατά της Ουγγαρίας σε σχέση με την νομοθεσία που ποινικοποιεί τη ΜΚΟ και την εργασία τους για τη στήριξη του ασύλου και που ε, δεν συνάδει το δίκαιο αυτό με το δίκαιο της Ένωσης. Δεν είναι συμβατό. Αυτή η υπόθεση είναι τώρα λοιπόν στο δικαστήριο. Το Δεκέμβριο του 2018 η Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου Ευρώπης είχε πει ότι ειδικό φόρος για τη μετανάστευση και η σχετική απόφαση παρεμβαίνει αδικαιολόγητα στην ελευθερία ε, δικαίου και έκφρασης ε, με αποτρεπτικό εφέ όσον αφορά τα άτομα που θέλουν να υπερασπιστούν το δικαίωμα ασύλου και τους, ε, συγγνώμη, τους, ε, το δικαίωμα να μπορούν να προσφέρουν οι ιδιώτες της εν λόγω ΜΚΕ. Ότι όλα αυτά δηλαδή είναι παράνομα για την περάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκε ότι αυτές οι διατάξεις θα πρέπει να καταργηθούν. Μπορείτε να μας διασυμβεβαιώσετε ότι αυτό το σημαντικό θέμα για τη δράση των ΜΚΟ που συζητήθηκε δεόντως στη διάρκεια των ακροάσεων υπό το άρθρο 7, ότι τελικά η Ουγγαρία συμμορφώνεται προς αυτά τα πορίσματα και τις αποφάσεις. Ε, κυρία θα ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου για το ότι το θέμα αυτό προγραμματίστηκε τέτοια ώρα. Α, λοιπόν που ξεκινώ με αυτό και ξέρω ότι δεν σχετίζεται, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει προγραμματιστεί εγκαίρως. Ε, και κάποια ώρα που θα ήταν και εδώ οι ευρωβουλευτές. Τώρα όμως θα μιλήσω ουγγρικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ με τους ε, συναδέλφους ε, να πω το εξής. Πριν από ένα χρόνο αποφασίσαμε, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με το ΕΛΚ, ε, στο οποίο εντάστηκε το Φίντες, να προστατεύσουν την ε, Ουγγαρία από την καταστροφή. Γι' αυτό ξεκίνησε και η διαδικασία του άρθρου 7. Θέλανε ακριβώς να σταματήσει η χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για διαφθορά, αλλά τίποτα δεν ε, σταματάει τον Όρμπαν, ούτε καν η αναστολή συμμετοχή του κόμματό του στο ΕΛΚ. Και ακόμα και τώρα, παρά το ότι έχασαν στις δημοτικές εκλογές, συνεχίζουν να διαλύουν το κράτος δικαίου. Και τώρα ακριβώς ε, έχουν μία νέα πρόταση που δίνει ακόμα ισχυρότερο έλεγχο ε, στην κυβέρνηση επί των δικαστηρίων. Και τώρα πλέον αποφασίζουν αυτοί για διάφορα δύσκολα ζητήματα. Υπάρχουν διάφορες ατασταλίες. Ε, τεράστια ποσά έπρεπε να επιστραφούν ε, πλέον από την Ουγγαρία. Λοιπόν, τι θα γίνει, μπορούμε να κάνουμε κάτι με το άρθρο 7 ή πρέπει να γράψουμε νέα έκθεση που θα περιλαμβάνει και αυτά τα γεγονότα. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί συναδελφοί εδώ πέρα που ασχολούνται με το θέμα του κράτους δικαίου και θέλουν να προστατεύσουν ακριβώς ε, την δημοκρατία. Είναι ευρωπαϊκό το ζήτημα. Πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά τη διαδικασία του άρθρου 7. Λοιπόν, δεν θέλω να τιμωρήσω την πατρίδα μου, όχι, θέλω διαδικασίες, θέλω η χώρα μου να είναι δημοκρατική και να προστατεύσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες. Οπότε θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι όλα αυτά αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο και μπορείτε να τα δείτε. Μάλιστα δεν βλέπω άλλους βουλευτές. Να επιτρέψατε μου ως ε, πρόεδρος ε, να αντιδράσω έτσι αυθόρμητα σε αυτήν την κριτική που την έχω ακούσει συχνά όσον αφορά την προσέλευση ε, πέμπτη στην Επιτροπή μας γιατί αυτό είναι αυτοκριτική. Δεν είναι κάτι το οποίο θα δέχομαι εγώ στο Προεδρείο, αλλά κάτω στα έδρανα. Γιατί πιστέψτε με, συχνά εγώ περιγράφω την ΛΥΜΠΕ ως την πιο πολύ άσχολη επιτροπή. Λοιπόν, η συνεδριά μας είναι κάθε εβδομάδα. Κάνουμε τις πιο πολλές ψηφοφορίες. 24% των ψηφοφοριών στην Ολομέλεια αφορά τη δική μας Επιτροπή. Δεν υπάρχει και κάποια Ολομέλεια στην οποία δεν πληρώνω το τίμημα πολιτικά και προσωπικά του να μην πηγαίνω στην Ολομέλεια και σε πολλά ζητήματα που με αφορούν γιατί προεδρεύω. Αλλά τι κάνουμε. Φορτώνουμε το πρόγραμμά μας και εντωμεταξύ σήμερα δεν κάναμε ε, τίποτα άλλο παρά μόνο συζήτηση για την κατάσταση των μεταναστών που επιστρέφονται στη Λιβύη. η ανθρωπιστική κατάσταση των κέντρων ε, στη Λιβύη. Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Επιχειρήσεις Σόφια. Όλο το πρωί. Με πολύ χαμηλή προσέλευση. λύπη μου. Πραγματικά δηλαδή. Ε, εγώ ε, απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Και τώρα πάλι άρθρο 7 που το ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τόσο χαμηλή προσέλευση το συζητάμε. Πρέπει να το ξανασκεφτούμε λοιπόν. Και να δούμε λογικά τη δουλειά της Επιτροπής μας. Γιατί ε, συνεχώς βάζουμε πράγματα στην ημερήσια διάταξη επιτροπής μας και οι βουλευτέ μα δείχνουν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν ε, στη δουλειά που οι ίδιοι παράγουν. Οπότε, ε, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε και να πούμε ε, εντάξει, οκ, okay, ε, ας το σκεφτούμε. Ας ηρεμήσουμε λίγο. Αλλιώ συμβαίνει πράγματι ότι έχουμε τόσο σημαντικά θέματα στη μερική διάταξη με χαμηλή προσέλευση γιατί ο κόσμος είναι αλλού ή επιστρέφουν στη χώρα τους, Όπω συνήθω συμβαίνει πέμπτη απόγευμα. Τώρα λοιπόν έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε σήμερα και όπως είπα εξ αρχής, το να ε, ε, βόμαστε τις κοινέ αρχές και το κράτος δικαίου είναι κρίσιμο για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το λόγο είναι μία από τις προτεραιότητες που αποφάσισε να θέσει η Φινλανδική Προεδρία όταν ε, αποφάσισε για το πρόγραμμα στη διάρκεια της Προεδρίας. Προχωρήσαμε σε τέσσερα διαφορετικά μονοπάτια όταν ξεκινήσαμε. Καταρχάς, ο κανόνας του διαλόγου είναι πολύ σημαντικός. Θέλουμε να το αναπτύξουμε ως ετήσια υπόθεση και να μην εστιάζουμε μόνο σε κάποια κρατημέλη, αλλά να εξετάζουμε την κατάσταση σε ολόκληρη την Ευρώπη και να έχουμε και έγκαιρη προειδοποίηση και εφόσον δούμε ότι κάτι ε, πάει, αρχίζει να πηγαίνει στραβά. Αυτό είναι κάτι που λοιπόν που θα θέλαμε να συνεχίσουμε στο τελευταίο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ε, στα απορίσματα του Συμβουλίου νομίζω υπάρχει μια πολύ καλή βάση για την εργασία μας για αυτό το θέμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο μέσα στην εργαλειοθήκη. Το δεύτερο στοιχείο που αναφέρθηκε από την κυρία Ισίρ είναι οι ε, ε, όροι στο PDP, η αιρεσιμότητα. Και αυτό είναι ένας άλλος δρόμος στον οποίο δουλεύουμε. Ε, τώρα ο, ολοκληρώνουμε το διαπραγματευτικό κουτί για το PDP που θα συζητηθεί στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκέμβριο. Και ο κανόνας ε, της ερεσιμότητας είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πιθανότατα θα αποφασιστεί στα τελευταία στάδια της διαπραγμάτευσης ανάμεσα στους ε, ηγέτες μας. Έπειτα, Είχαμε αυτό το άρθρο 7 για τη σχετική διαδικασία που συνεχίζεται. Ξεκίνησε αυτή η ακρόαση με την Ουγγαρία επειδή, όπως είπα, θεωρήσαμε πως ε, είχαν περάσει χρόνια από τότε που το, μάλλον ένας χρόνος από τότε που έκανε το ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οπότε έπρεπε να γίνει η ακρόαση και έπειτα ε, η τέταρτη αναζήτηση ήταν εκτό των θεσμών και ήταν η πρωτοβουλία που να, ε, πρόταξαν η Γερμανία και το Βέλγιο, δηλαδή η... Ε, επιδόσεις και η σύγκριση μεταξύ των ε, ομολόγων. Και αυτό το ε, παρακολουθούμε στενά σε συνεργασία με αυτές τις δύο χώρες. Πολύ ρώτησατε ποιος τρόπος είναι ο καλός για να προχωρήσουμε. Και βεβαίως ο τρόπος που θα προχωρήσουμε εξαρτάται από την επόμενη Προεδρία και τα κράτη-μέλη όλα που πρέπει να αποφασίσουν ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε. Τώρα έχουμε αποφασίσει να γίνει αυτή η δεύτερη ακρόαση για την ε, Ουγγαρία στο επόμενο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και είναι πολύ σημαντικό. Είμαι ικανοποιημένη που δώσατε πολλές ιδέες και τροφή προσκέψη και για την Προεδρία στην προετοιμασία της ακρόασης μαζί με τα άλλα κρατημέλη. Η κορεπέρ της επόμενης εβδομάδας είναι αυτή που θα αποφασίσει ποια θα είναι τα θέματα της επόμενης ακρόασης και βεβαίως είμαστε πρόθυμοι να έχουμε την συμβολή σας, να τη δώσουμε στην Προεδρία και αυτό μας βοηθάει όταν αποφασίζουμε από κοινού με τα κράτη-μέλη τα θέματα να τα δώσουμε δηλαδή και στην κροτική προεδρία. Αλλά βέβαια υπάρχουν πολλά θέματα και αυτή η ακρόαση, αυτό δηλαδή που κάνουμε τώρα, θα πρέπει να είναι μέσα στο πλαίσιο της έκθεσης, της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συζητήθηκαν ε, και οι νέες εξελίξεις ε, και βεβαίως αυτές οι νέες εξελίξεις θα μπορούσαν να συζητηθούν ανάμεσα στα θέματα που αναγράφονται στην έκθεση. Η έκθεση είναι πολύ εμπεριστατωμένη και πιστεύω πως ε, τα περισσότερα ζητήματα τα περιλαμβάνει, αυτά που αναφέρατε δηλαδή. Και Αν θέλετε να έχετε περισσότερες λεπτομέρειες για την επόμενη ακρόαση, δεν μπορώ να σας πω τώρα τίποτα, γιατί δεν έχει αποφασιστεί στην Κορεπέρ. Ε, θα πρέπει να φέρουμε τα κράτη-μέλη λοιπόν στο ίδιο τραπέζι και μετά να αποφασίσουμε τα θέματα και φυσικά, όπως είπα, είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε και τις δικές σας ιδέες. Τέλος, όσον αφορά το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου και ξέρω ότι έχει υπάρξει με πολύ κριτική παραπονά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει προσκληθεί στα συμβούλια όταν συζητάμε δηλαδή τα θέματα της διαδικασίας του άρθρου 7 αλλά το Συμβούλιο είναι της άποψης ότι το χρειάζεται να υπάρχει αγαστή συνεργασία με το Κοινοβούλιο, βεβαίως, αλλά το θέμα του πώς θα συμμετέχει το Κοινοβούλιο συζητήθηκε στο Συμβούλιο όταν ε, διαπραγματευτήκαμε τις στάνταρ ε, διατυπώσεις και τα κάτι μέλη επέλεξαν η Προεδρία να είναι σε επαφή με το Κοινοβούλιο και μετά να ενημερώνει το Συμβούλιο για τα σχόλια που έκανε το Ευρωκοινοβούλιο. Και ένα αυτός ένας από τους λόγους για τους οποίους βρίσκομαι σήμερα εδώ. Και αυτό πρέπει πολύ προσεκτικά να τα ε, μελετήσουμε για να ενημερώσουμε το Συμβούλιο στις αρχές ε, ε, του επόμενου χρόνου για όλες αυτές τις διατυπώσεις. Επίσης τώρα ως Προεδρία προβληματιζόμαστε για το πώς θα οργανώσουμε τη συνεργασία μαζί σας στο υπόλοιπο της Προεδρίας μας και θα επανέλθουμε σε αυτό το χρόνο. Αλλά ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει εδώ. Θα επανέλθουμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας που ήταν εξαιρετικά χρήσιμα για μας επειδή τώρα προετοιμάζουμε το επόμενο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ. Εντάξει, αρκετά είναι, δεν έχουμε άλλα σχόλια. Αρκετά είναι όλα αυτά που ακούσαμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και νομίζω ότι σύντομα θα πρέπει να ε, εξορθολογήσουμε το φόρτο εργασίας της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ όλους.